Καλησπέρα σε όλους σας και στην αίθουσα εδώ και στο Βερολίνο και καλώς ήρθατε στην συνεδρίασή μας και χαιρετώ και τον κύριο Χίνσκερτ, τον επίσης κύριο Πρόεδρο. Μπορούμε νομίζω να ανταλλάξουμε λίγα λόγια για να δούμε αν ακούγόμαστε καλά πριν περάσουμε στην ε, συνεδρίαση. Οπότε ευχαρίστω να σας δώσω τον λόγο για να καλωσορίσετε και τους βουλευτές εδώ πέρα. Σας ε, χαιρετώ, ελπίζουμε, χαιρόμαστε κι εμείς ιδιαίτερα, ελπίζω να έχουμε μια επικοδομητική συζήτηση και να ε, μας φέρει και πιο κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εμείς ε, σας βλέπουμε μια χαρά. πρέπει βεβαίως να μιλάει ο ένας μετά τον άλλον. Δεν είναι τόσο άμεση η συνομιλία μας, αλλά ξέρω πως έχετε πολλές ερωτήσεις για μας. Πρώτα απ' όλα να σας πω, γιατί βεβαίως αυτά μεταδίδονται και στο διαδίκτυο και θα το βλέπουν παντού. Οπότε πρόκειται για την πιλωτική εφαρμογή μιας νέας ε, τεχνολογίας από πλευράς ε, του Κοινοβουλίου για τηλεδιασκέψεις υψηλής ευκρίνειας και νομίζω πως είμαστε η πρώτη επιτροπή που συνεργαζόμαστε με άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή Οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ του συναδέλφου ε, της Γερμανικής Ομοσπονδιακής ε, Βουλή που συμφώνησαν σε αυτό. Οπότε, για το πώς ε, θα κυλήσουν πρακτικά τα πράγματα. Εμείς εργαζόμαστε στην συνήθη αίθουσά μας, θα δείτε πως είναι αρκετά μεγάλη και οι συνάδελφοι είναι κανονικά στις αίθουσές τους και βεβαίως όταν ανάβει το μικρόφωνο τους τους βλέπετε πιο κοντά. Οπότε θα έχετε άμεση αντίδραση από τα μέλη μας εδώ πέρα. Και θα γίνει έτσι μια συζήτηση. Όπως ξέρετε η αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων είναι μια πολιτική κλειδί όσον αφορά την Επιτροπή μας για τις αρμοδιότητες μας ε, στον τομέα της εσωτερικής αγοράς και προστασίας των καταναλωτών. Η Κομισιόν ε, επεξεργάζεται μια αλλαγή αυτής της πρότασης, την οποία βεβαίως ε, αναμένουμε και για να προετοιμαστεί η πολιτική μας θέση ε, θα συντάξουμε μία έκθεση που θα κοιτάει και την εφαρμογή της υφιστάμενης οδηγίας και το πώς θέλουμε να αλλάξει και θα ακούσετε σε λίγο την εισηγήτριά μας, την κυρία Έμα Μακλάρκιν και αναμένουμε η Κομισιόν να μας στείλει μια νομοθετική πρόταση γύρω στο Δεκέμβριο νομίζω. Η κυρία Μακλάρκιν θα μας πει λίγο για το πότε θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Οπότε θέλουμε και τις απόψεις σας καθώς θα γίνει αυτή η συζήτηση. Αυτά από μένα ως εισαγωγή. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Χίντσκεν, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής στην Ομοσπονδιακή Βουλή για να κάνει μια εισαγωγή. Μετά η κυρία Μακλάρκεν θα κάνει μια εισαγωγή και νομίζω πως μετά κύριε Πρόεδρε και οι δύο μας έχουμε ένα κατάλογο και ελπίζω προς το τέλος να υπάρχει λίγος χρόνος για μια συζήτηση ελεύθερη αρκεί βεβαίως να τηρήσουν όλοι οι συνάδελφοι το χρόνο ομιλίας και οι συνάδελφοί μου εδώ πέρα ούτως ή άλλως θα βλέπουν το ρολόι και είμαι σίγουρος πως και εσείς θα χρονομετράτε όπως κάνουν όλοι οι πρόεδροι. Οπότε σας προσκαλώ να απευθύνετε και σε ένα χαιρετισμό σε μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χάρμπορ. Ως εισαγωγή να πω πως ε, εμείς ε, στη γερμανική πλευρά Είμαστε βεβαίως ούτως ή άλλως η Επιτροπή για την Οικονομία και την Τεχνολογία, οπότε χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την πιλωτική αυτή εφαρμογή με την οποία συζητάμε σήμερα. Έρχομαι αμέσω στο θέμα μας για να μην σπαταλούμε χρόνο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το ότι αγαπητοί συνάδελφοι της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Εσωτερική Αγορά και οι δικοί μας οι συνάδελφοι θα μπορούν να συζητήσουν αυτό το θέμα. Γιατί η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην Ευρώπη έχει αποφασιστική σημασία έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε με βέλτιστο τρόπο το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό στην Ευρώπη και να βελτιωθεί η κινητικότητα στην Ευρώπη. Οπότε η ε, επεξεργασία αυτής της ε, οδηγίας ε, έχει ιδιαίτερη σημασία. Χαιρόμαστε για το ότι η Επιτροπή Αγοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασχολείται με αυτό το θέμα και σας ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία για αυτή τη βιντεοδιάσκεψη. Το σχέδιο έκθεσης ε, της ε, κυρίας ε, Έμας Μακλάρκιν το διαβάσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Η Γερμανία υποστήριξε εξ αρχής το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας επαγγελματικών προσόντων. Τα δε προηγούμενα έτη έχουμε ήδη επιτύχει πολλά. Επίσης, η επεξεργασία αυτής της ε, οδηγίας μας δίνει τη μεγάλη ευκαιρία να καταστήσουμε αυτή τη διαδικασία αναγνώριση ακόμη απλούστερη, πιο διαφανή και φιλική προς το χρήστη. Και χαιρετίζουμε από τη γερμανική πλευρά το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πράσινη βίβλο της συμπεριέλαβε πάρα πολλές γερμανικές προτάσεις πολλά από τα μέτρα τα οποία προτείνονται εδώ πέρα είναι κατά την άποψή μας ενδεδειγμένα έτσι ώστε να επιτρέψουν στους πολίτες να εργαστούν σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα χωρίς να αμφισβητηθεί καθόλου το υψηλό επίπεδο ποιότητας. Και με τη σημερινή βιντεοδιάσκεψη έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να συζητήσουμε το ποιε είναι οι ανάγκε για αλλαγές που χρειάζονται. Υπενθυμίζω παραδείγματο χάρη το ζήτημα της επαγγελματικής ταυτότητας για την ε, εισαγωγή της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη το Φεβρουάριο του 2009 είχε εκφραστεί θετικά. Μέσω μιας τέτοιας ταυτότητας που θα εκδίδεται από το κράτος μέλος προέλευσης θα μπορούν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή υποδοχής να έχουν μια υποστήριξη όσον αφορά την εξέταση των επαγγελματικών προσόντων. Ενδιαφέρον επίσης είναι το ζήτημα το για ποια άλλα επαγγέλματα θα μπορούσαμε να ορίσουμε κάποιες ελάχιστες εκπαιδευτικές προδιαγραφές και άρα να έχουμε την αυτόματη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και σε αυτά. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει συζήτηση και για το θέμα της κατάργησης των διαφόρων φάσεων των απόκτησης των προσόντων. Πρέπει να το δούμε αυτό πάρα πολύ σοβαρά. Ήμουν σύντομος, νομίζω πως υπάρχει ήδη και αρκετή εμπειρία και από τη δικιά μας την ε, πλευρά. Θα προσπαθήσω λοιπόν να ακουστούν όλοι οι συνάδελφοι και Οπωσδήποτε αναμένουμε το τι έχετε να μας πείτε και εσείς από τις Βρυξέλλες για να οδηγηθούμε σε μια λογική και επιτυχημένη λύση. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη συνεργασία. Ευχαριστώ που θέσατε ευθέως τις ανησυχίες που έχουμε και πολλοί από εμάς. Θα δώσω το λόγο στη Μακλάκη, την εισηγήτριά μας τέσσερα λεπτά για να μπορέσει να κάνει την εισαγωγική της παρουσίαση και μετά θα σας ξαναδώσω το λόγο, Πρόεδρε, για να παρουσιάσετε τον πρώτο σας συζητητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Μεγάλη χαρά για μένα που παίρνω μέρος σε αυτή την συνάντηση σήμερα. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και του Bundestag. Είμαι σίγουρος ότι η ανταλλαγή απόψεων θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Είναι η πρώτη φορά που είμαι εισηγήτρια από τότε που εξελέγην. Ενδιαφέρομαι για το θέμα εδώ και ένα χρόνο όταν ήμουν εισηγήτρια επιγνωμοδοτήσεως για τα θέματα των επαγγελμάτων υγείας και για τη δυνατότητα των επαγγελματιών του τομέα της υγείας να λειτουργούν διασανοριακά. Ε, όχι μόνο είναι κρίσιμη η παρούσα οδηγία για την ανάπτυξη αλλά και για την κινητικότητα των πολιτών και για τη διασφάλιση των ασθενών και γενικότερα των πολιτών. Νομίζω ότι η μελλοντική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απασχολεί πάρα πολλές επαγγελματικές κατηγορίες και όλοι συμφωνούν στο ότι οι επαγγελματίες στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιμένουν να δώσουμε τις σωστές προτάσεις. Οι επαγγελματίες αυτοί προσπαθούν να βοηθήσουν τους πολίτες να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής και θέλουν να λειτουργήσουν και να προσφέρουν και στην ενιαία αγορά. Πρέπει να τους δώσουμε αυτή τη δυνατότητα. Θέλουν να υπάρξει ένα streamlining των διαφόρων συστημάτων για την ελεύθερη διακίνηση και θέλουν και κανόνες για τη διασφάλιση της ποιότητας θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην επιβαρύνουμε με απαράδεκτα κόστη και με γραφειοκρατικές δυσκολίες τους σωστούς επαγγελματίες. Το Green Paper της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η διαβούλευση που, που διεξήχθη είναι πλέον διαθέσιμες. Υπήρξαν πάρα πολλές ανταποκρίσεις από τα 27 κράτη και τις 27 δημόσιες αρχές, επαγγελματικά σώματα, κυβερνήσεις κτλ. Λοιπόν, αναγνωρίστηκε ότι το σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης είναι ρεαλιστικό και αποτελεσματικό, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς στους οποίους θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές. Έχοντας αναθεωρήσει όλα αυτά τα συστήματα, μπορώ να καταλήξω στο ότι η δυσαρέσκεια στη σημερινή κατάσταση εξηγείται από την έλλειψη εμπιστοσύνη στο υπάρχον σύστημα. Τα κράτη-μέλη και οι αρμόδιες αρχές παραπονούνται για περιορισμένες πληροφορίες και οι επαγγελματίες παραπονούνται για την έλλειψη στην Ευρώπη του 21ου αιώνα η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της υγείας διασύνοριακά είναι μια απόδειξη της ενεργής λειτουργίας της, ελεύθερης, της εσωτερικής αγοράς. Κάτι το οποίο λοιπόν πρέπει να βοηθήσει την κινητικότητα των επαγγελματιών μέσω της άμεσης και εύκολης αναγνώρισης των επαγγελματικών τους ικανοτήτων μέσα από τα συστήματα που λειτουργούν στις διάφορες χώρες και διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών για την προστασία των ασθενών. Εγώ προσπάθησα όλους αυτούς τους στόχους να τους λάβω υπόψη. Θέλω εγώ η οδηγία αυτή να λειτουργήσει καλύτερα για τους πολίτες και θα πρέπει να δημοσιεύεται online η δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων. Ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξυγχρονίσει κάποιες από τις προβλέψεις της συγκεκριμένης οδηγίας που είναι 30 σχεδόν ετών και απαιτούν νέα διατύπωση αλλάζοντας επίσης τις ελάχιστες επαγγελματικές απαιτήσει ε, για να υπάρχει ανταπόκριση στις σημερινές απαιτήσει και εντάσσοντας και την ιδέα της συνεχούς κατάρτισης στην παρούσα διαδικασία και ορίζοντας ότι τα επαγγέλματα αυτά παραμένουν σε ένα χώρο ο οποίος είναι ελεγχόμενος επαγγελματικών δραστηριοτήτων ελεγχόμενων διασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ελευθερία της λειτουργίας της αγοράς. Και οι προτάσεις για την επαγγελματική κάρτα ή επαγγελματική ταυτότητα δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικές θα πρέπει όλα αυτά να συνδεθούν με το σύστημα ενημέρωση τη εσωτερική αγορά, όπως επίσης και με το σύστημα έγκαιρη προειδοποίηση στην περίπτωση κατά την οποία έχουν υποστεί κάποιοι επαγγελματίε κυρώσει στις συγκεκριμένες χώρες προέλευση. Υπάρχει και το θέμα των γλωσσικών ικανοτήτων, είναι κάτι το οποίο όμω θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω η μερική πρόσβαση σε αγορές είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω διαβουλεύσεων. Οι διαβουλεύσεις μέχρι τώρα έχουν δείξει ότι δεν θα ήθελαν οι ιδέες αυτές να ενταχθούν στη συγκεκριμένη πρόταση οδηγίας. Θεωρούν ότι υπάρχουν εδώ πάρα πολλές παγίδες οι οποίες δεν μπορεί να καλυφθούν. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει περαιτέρω έρευνα των προτάσεων αυτής, αυτών πριν καταλήξουμε στις πιθανώς συνέπειες οι οποίες μπορεί να προκληθούν. Θέλω λοιπόν να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων για το πώς η οδηγία αυτή μπορεί να καταστεί καλύτερη και για την κοινότητα και για τους επαγγελματίες. Θα δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στον Συμπρόεδρο να μας πει ποιος θα είναι ο πρώτος του ομιλητής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την τοποθέτηση της εισηγήτριας και θα δώσω τον λόγο στους εκπροσώπους των διαφόρων κοινοβουλευτικών ομάδων. Πρώτος, πρώτη, έχει τον λόγο η κυρία Σιόν μέλος της ε, κοινοβουλευτικής ομάδας του Τσεντεού Τσέσου. Κυρία Σόεν, έχετε τον λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Bundestag, σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε να τοποθετηθούμε και για την οργάνωση αυτής της ανταλλαγής, γιατί εξυπηρετεί την καλύτερη συνεργασία των κοινοβουλίων. Βεβαίως το θέμα μας είναι η εφαρμογή της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα που αποτελεί βεβαίως προϊόν της κοινή μας θέλησης να διαμορφωθεί σωστά η ελευθερία διακίνησης των ε, πολιτών. Κατά την ε, επεξεργασία αυτής της οδηγίας η Γερμανία έχει καταθέσει ήδη πάρα πολλές ε, προτάσεις, ε, τις οποίες υιοθέτησε η Κομισιόν και γι' αυτό την ευχαριστούμε. Για λόγους ε, συντομίας, επειδή έχω μόνο δύο λεπτά, θα περιοριστώ μόνο σε τέσσερα σημεία για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και καλύτερα. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε αυτή την ε, μερική αναγνώριση των προσόντων αρκετά επικριτικά γιατί εμείς έχουμε ένα διαφορετικό σύστημα και ειδικά το σύστημα της διπλής εκπαίδευσης που έχουμε εμείς διακινδυνεύει και έχει αποδειχθεί πολύ επιτυχές στην ε, Γερμανία και στο να μειώσει την ε, ανεργία των νέων. Δεύτερον, το ότι αυξάνονται τα κριτήρια εισαγωγή ε, στα επαγγέλματα υγείας είναι κάτι το οποίο βλέπουμε επικριτικά καθώς νομίζουμε πως μετά από χρόνια ε, σπουδών μπορούν να επιδείξουν μια υψηλή ποιότητα επαγγελματίες υγείας και δεν θεωρούν πως υπάρχει κάποια ανάγκη αλλαγής. Το άλλο το οποίο βλέπουμε κάπως επικριτικά είναι οι λεγόμενες ταυτότητες ε, του επαγγελματία, οι professional cards. Το χαιρετίζουμε οπωσδήποτε, αλλά θα πρέπει να πούμε πως η αναγνώριση των προσόντων είναι κάτι το οποίο παραμένει υπόθεση της χώρας υποδοχής. Βεβαίως η κάρτα αυτή μπορεί να αποτελέσει μια βάση, αλλά δεν θα πρέπει να προδικάζει το αποτέλεσμα. Και τέλος όσον αφορά την μεταρρύθμιση αυτόματης πλατφόρμας για την ε, αμοιβαία αναγνώριση. Θεωρούμε σωστό το... την πρόταση για να μειωθεί η ελάχιστη αυτή παρουσία κρατών μελών που απαιτείται στον αριθμό των 9 ε, μεν σωστή, αλλά υπάρχει εδώ πέρα ο κίνδυνος του κατακαιρματισμού. Σας ευχαριστούμε λοιπόν εκ των προτέρων για την συνεργασία μας που θα είναι προς το συμφέρον των πολιτών και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Έχετε λοιπόν τον λόγο εσείς πάλι κύριε Χάρμπορ. Ευχαριστώ. Ναι, διαμορφώνουμε μια καλή εικόνα και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι υπάρχει διερμηνία σε όλες τις επίσημες γλώσσες και ευχαριστώ και τους διερμηνείς Γι' αυτό θα δώσω τώρα το λόγο στους και οδησηγητές, όπως λέμε, από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Η κυρία Μακλάρκιν είναι από τους Ευρωπαίους Συντηρητικού και Μεταρρυθμιστές. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Αλεγκρίπ Κόνσταν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους από το Bundestag για τη συμμετοχή σε αυτή την τηλεδιάσκεψη που στόχο έχει την στενότερη συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που μα είναι ιδιαίτερα προσφυλή. Επευκαιρία αυτή αυτής της ανταλλαγής απόψεων και συνεχίζοντα το φόρουμ για την εσωτερική αγορά που έγινε πριν από λίγε μέρε στην Κρακοβία, είχαμε τότε την ευκαιρία να συζητήσουμε και με επαγγελματίε, με εκπροσώπου Κοινωνία των πολιτών, με ε, βουλευτέ διοικητικού από διάφορε χώρε. και γνωρίζουμε ότι στη Γερμανία υπάρχουν πολλές προτάσεις και μεγάλες ανησυχίες για τον εξυγχρονισμό της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Ε, και οι ανησυχίες αυτές αφορούν την ε, μερική πρόσβαση, την παροχή υπηρεσιών, την προορατική προειδοποίηση και την επαγγελματική ταυτότητα. Αυτά είναι μερικά από τα πιο ευαίσθητα σημεία και τα πιο σημαντικά, πιο σημαντικές προκλήσεις αυτής της ε, αναθεώρησης της ε, σχετικής νομοθεσίας. Και η έκθεση που θα ψηφίσουμε σε λίγο στην Επιτροπή ΜΚΟ λαμβάνει υπόψη και αυτές τις ανησυχίες και αυτές τις προτάσεις της Γερμανικής Βουλής. Και ε, ελπίζω ότι θα στηρίξουμε και σημαντικά σχέδια που είναι προσφυλή και στα Εθνικά Κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να διευκολύνουμε την κινητικότητα των επαγγελματιών. Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων είναι μία από τι 50 προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πράξη για την εσωτερική αγορά, που ήταν ένα από του σημαντικότερου 12 άξονε ανάπτυξη, όπω επισήμανε ο Επίτροπο Μπαρνιέ. Και εν ώψη τη αναθεώρηση ε, τη σχετική νομοθεσία ε, που θα κάνουμε τον επόμενο χρόνο, θα ήθελα να αναφερθώ στο ιδιαίτερο θέμα τη ε, Ευρωπαϊκή Επαγγελματική ταυτότητα. Κατά τη γνώμη μου αυτή η ταυτότητα, η επαγγελματική ταυτότητα θα, πρέ... θα μπορούσε να είναι συγκεκριμένο εργαλείο τη κινητικότητα των επαγγελματιών. Θα απλουστεύσει την κατάσταση, αλλά θα κάνει και πιο αποτελεσματική την κατάσταση και για τους επαγγελματίες αλλά και για τις αρμόδιες αρχές και τα κράτη-μέλη. Γιατί θέλουμε μια Ευρώπη των πολιτών και από αυτή την άποψη θα έχουμε πολύ σημαντική και απτή πρόοδο που την περιμένουν και οι συμπολίτε μας. Φυσικά υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για τη θέσπιση αυτή τη επαγγελματική ταυτότητα από τεχνική άποψη, τι είδου ταυτότητα θέλουμε, τη βάση δεδομένων, πώ θα τα εξυγχρονίσουμε, πώ θα τα ενημερώσουμε. Υπάρχουν νομικά θέματα, προστασία δεδομένων, οικονομικά ζητήματα, το κόστο. Θα πρέπει να διαλευκάνουμε όλα αυτά τα θέματα και τα προσεγγίζουμε στην έκθεση τη κυρία Μακλάρκιν και από αυτήν την άποψη περιμένουμε τι δικέ σα προτάσει. Το σημαντικό πάντως είναι οι ταυτότητες αυτές να μην είναι γενικευμένες αλλά οικειοθελείς και να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία ορισμένων επαγγελμάτων, για παράδειγμα των μηχανικών στη Γερμανία, που ήδη εφαρμόζουν μια τέτοια επαγγελματική κάρτα ή επαγγελματική ταυτότητα. Πάντω, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι και το ίδιο και οι επαγγελματίε μα και σα ευχαριστώ για τι προτάσει σα στο συγκεκριμένο αυτό θέμα. Uh, thank you very much, Mrs. Ευχαριστούμε κύριε Λεγκρίπ. Κύριε Πρόεδρε Χίσκινγκ, ε, παρέλειψα να καλωσορίσω και τον ε, υπεύθυνο της, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Αρμόδια Γενική Διεύθυνση, τον κύριο Γιώργαν Τίτζη, που είναι και ο αρμόδιος ε, για τη σχετική πρόταση και είναι παρόν εδώ και θα παρακολουθήσει τη συζήτηση. Και αν μας μείνει χρόνο στο τέλος, θα του δώσω το λόγο για μερικά σχόλια είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε. Θα σας δώσω το λόγο τώρα για να μας ορίσετε τον επόμενο μιλητή. Ε, Ευχαριστώ. Εφόσον το επιτρέπει ο χρόνος, θέλουμε να κάνουμε όσο περισσότερα μπορούμε. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον συνάλφο τον Κράους Μπάρτελ, που είναι πρόσωπος για αυτά τα θέματα των social δημοκρατών. Κύριε Μπάρτλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και καλημέρα σε όλους. Εμείς συμφωνούμε με τους στόχους ε, του σχεδίου της νέας ε, οδηγίας, αλλά θεωρούμε πως οι προτάσεις ε, εν μέρη μόνο αντίκνεται για αυτούς τους στόχους, οπότε ελπίζουμε η διάσκεψη αυτή να μην αποτελεί μόνο μια τεχνική ε, άσκηση αλλά να συνεισφέρει και στην διαδικασία αναθεώρησης οδηγίας. Να πω πρώτα απ' όλα πως προφανώς υπάρχει μια ευρεία συμφωνία για τα ζητήματα αυτά μεταξύ των μεγάλων κομμάτων. Να αναφέρω πως ε, τα τέσσερα σημεία τα οποία ανέφερε στην Αλφοσέν μας βρίσκουν και εμάς ε, σύμφωνους. Επίσης να παρατηρήσω πως είχαμε μία αντιπαράθεση για την οδηγία υπηρεσιών και εμείς θεωρούμε πως η οδηγία επαγγελματικών προσόντων δεν πρέπει τώρα να χρησιμοποιηθεί για να έρθουν πάλι, να έρθει ξανά η αρχή της χώρας προέλευσης από την πίσω πόρτα. Γι' αυτό ο τονισμός ορισμένων μεμονωμένων περιπτώσεων όπως ε, παραδείγματος χάρη ο συνοδός μιας εκδρομής δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για να αλλάξει ολόκληρο το σύστημα επαγγελματικών προσόντων. Αυτές είναι μεμονωμένες περιπτώσεις που δεν θα πρέπει να επηρεάζουν το συνολικό σύστημα. Δεύτερον, να τονίσω πως θεωρούμε λογική και την επαγγελματική ταυτότητα, αλλά δεν σημαίνει κάποιον αυτοματισμό και θα πρέπει να διατηρηθεί η διαδικασία αναγνώρισης ε, της ε, χώρας υποδοχή και θα πρέπει επίσης η κάρτα αυτή να περιέχει κάποια προσωπικά δεδομένα. Επίσης θα πρέπει να ε, διατηρήσουμε την συνολική προσέγγιση. Βλέπουμε πάρα πολύ επικριτικά την κατάτμιση αυτή των προσόντων και επίσης θέλουμε το σύστημα κατάταξης να μην γίνει ακόμη πιο πολύπλοκο. Γι' αυτό ζητάμε το σύστημα ακριβώς κατάταξης των επαγγελμάτων να είναι όσο το δυνατόν πιο απλό. Παραδείγματο χάρη να ακολουθεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων και επιπλέον υπενθυμίζουμε εδώ πέρα το πρόβλημα των γλωσσικών γνώσεων σε ορισμένα επαγγέλματα όπου από την πλευρά του χρήστη ή του καταναλωτή είναι απολύτως απαραίτητο αυτός ο οποίος παρέχει την υπηρεσία να γνωρίζει γλώσσες και βεβαίως εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική ρύθμιση. Το είπαν και οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ κύριε Μπάρτλ. Έχετε ξανά εσείς τον λόγο κύριε Χάρμπορ. Ευχαριστώ κύριε Μπέντετ Μενιού, είναι σκιώδη συζητήτρια για τους σοσιαλδημοκράτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα δώσει τη δική τη ε, συνεισφορά, συμμετοχή. Θα προσπαθήσω κύριε Πρόεδρε να σεβαστώ το χρόνο, λέει κυρία Βερνιό. Χαίρομαι για τις συζητήσεις αυτές με τα κοινοβούλια των κρατών μελών γιατί πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται μόνο μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και με τα κοινοβούλια των κρατών μελών που κατανοούν τα προβλήματα και συνεργάζονται μαζί μας τώρα. για την μεταρρύθμιση της συγκεκριμένης οδηγίας του 2005 συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι βασικό αυτό. Η οδηγία αυτή έχει δείξει ότι έχει πάρα πολλά κενά. Στα πλαίσια μιας κινητικότητας των εργαζομένων που αυξάνεται όλο και περισσότερο και θα συνεχίζει να αυξάνεται γιατί οι περισσότεροι νέοι γνωρίζουν ότι θα έχουν ανάγκη για την επαγγελματική του ζωή να πάνε και στο εξωτερικό. Κάποιο πρόβλημα τεχνικό υπάρχει και διακόπτει η κυρία Βερνιό. Μόνο τα γαλλικά ακούμε εμείς. Θα σας παρακαλέσω να... Α, τώρα, τώρα ακούμε κάποια γερμανικά. Να, τώρα σας ακούμε. Τώρα είναι όλα εντάξει. Moi qui suis particulièrement fatiguée aujourd'hui, mais ça fait rien, c'est du... Νιώθω μια κόπωση σήμερα, λυπάμαι. Τα ξαναλέω. Ίσως να υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα. Στα πλαίσια της οδηγίας αυτής άλλωστε ασχολούμεθα και με τα θέματα αυτοτεχνικά. Λοιπόν, θα ξαναπώ πάνω κάτω τα ίδια. Χαίρομαι που συνεργάζομαι με τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Πάντα υπερασπίστηκα τις αρμοδιότητές τους. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα δεν το προωθεί μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και το σύνολο των κοινοβουλίων που συνεργάζονται μαζί μας. Στα πλαίσια της αναθεώρησης της οδηγίας για τις επαγγελματικές ικανότητες 2005, συνειδητοποιήσαμε ότι έχει δείξει ότι έχει πάρα πολλά κενά. Γιατί η κινητικότητα των εργαζομένων αυξάνεται και θα συνεχίσει να αυξάνεται όταν βλέπουμε τις στατιστικές των νέων που θέλουν να πάνε να δουλέψουν στο εξωτερικό. Από ανάγκη πολλοί από αυτούς. Γι' αυτό λοιπόν οι νέοι Ευρωπαίοι επαγγελματίε πρέπει να μπορούν να κινούνται είναι σημαντικό για την εσωτερική αγορά, το έχουμε πει επανειλημμένα, για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας, την ανταγωνιστικότητα των χωρών μας. Θα πρέπει οι επαγγελματίες να νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, και γι' αυτό οι πολίτες, οι ασθενείς, οι πελάτες, όλοι θα πρέπει να νιώθουν και αυτοί ότι λειτουργούν σε ένα περιβάλλον ασφάλειας. Σημερίζομαι λοιπόν αυτά που είπε η συνάδελφος Λεγκρίπ, συμφωνώ και με αυτά που είπε και ο συνάδελφος του S5 και κανονικό είναι αυτό γιατί δεν μας χωρίζουν παρά λίγα σύνορα. Εγώ αντίθετα ε, για την επιμέρους ε, δυνατότητα εισόδου στην αγορά έχω προβλήματα. Και για τις γλωσσικές γνώσεις που δημιουργούν προβλήματα νομίζω ότι στην οδηγία αυτή για την αμοιβαία επαγγελματική αναγνώριση θα πρέπει να στοχεύσουμε σωστά τις μορφές ε, κατάρτισης. Δεν μιλάμε για αρχική κατάρτιση. Η συνεχής κατάρτιση δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες, η διαβίου κατάρτιση. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε στην δημιουργία της εκεί που δεν υπάρχει. Προφανώς και πρέπει να υπάρξει και γλωσσική κατάρτιση και για την κάρτα την επαγγελματική, την ταυτότητα την επαγγελματική, προφανώς είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι ιδιαίτερος χρήσιμο για την ευρωπαϊκή ταυτότητα, κάτι το οποίο θα δείξει ότι η ευρωπαϊκή αγορά δεν είναι μόνο η διακίνηση των προσώπων και των αγαθών, που έτσι και αλλιώς δεν είναι πολύ καλά ρυθμισμένη. Αλλά η κάρτα αυτή μπορεί να είναι πράγματι η βάση πάνω στην οποία θα δημιουργηθεί πλούτος που θα τον μοιράζονται όλοι οι πολίτες. Πρέπει σύντομα να έχουμε τα μέσα τα απαιτούμενα που να ευνοούν την κινητικότητα από τη μία, να ρυθμίζουν την κινητικότητα αυτή από την άλλη και να προσδίδουν και κριτήρια ασφαλείας στους επαγγελματίες και στους πελάτες τους. Ευχαριστώ Μπερναντέτ Βερνιό. Ε, δεν υπάρχουν προβλήματα μεταφορά της μετά της διευμηνίας στους Γερμανούς φίλους, τους ξαναδίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω και εγώ τον λόγο στην εκπρόσωπο των φιλελευθέρων, την κυρία Κλαουδία Μπέγκε, η οποία είναι η εισηγήτρια αυτών των θεμάτων ε, για τους ελεύθερους δημοκράτες. Κυρία Μπέγγελ, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Hello και bonjour στους ε, συναδέλφους της ε, Βρυξέλλες. Χαίρομαι που σήμερα έχω την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το ζήτημα εξ ονόματος της ομάδας μου και να σας πω πως η ομάδα του FDP των Φιλελευθέρων στην Ομοσπονδιακή Βουλή οπωσδήποτε χαιρετίζει την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας γιατί βεβαίως στόχο έχει να υπάρχει υψηλότερη, γρηγορότερη και καλύτερη κινητικότητα και ατόμων ε, και των προσόντων τους. Η έλλειψη των ε, εξειδικευμένων, ε, του εξειδικευμένου προσωπικού είναι ένα θέμα το οποίο βεβαίως μας απασχολεί συνεχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η οδηγία προσπαθεί να το αντιμετωπίσει. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει μια άμεση και εύκολη μεταφορά γνώσεως και ταλέντων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ως υπεύθυνη της ομάδας μου για τον τομέα των επιστημών να τονίσω εδώ πέρα τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις απαιτήσει αυτών των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις όμως ζητάνε και ένα διαφανές πλαίσιο σε σχέση με τις υπόλοιπες ε, πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης σας υπενθυμίζω εδώ πέρα τη διαδικασία της Κοπενχάγης που στόχο έχει την ολοκλήρωση ενός ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου. Οι περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της αμοιβαίας αναγνώριση επαγγελματικών προσώπων... είναι πάρα πολύ, ε, πάρα πολύ Δεν θα πρέπει όμως να έχουν ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο μέλλον ένα βουνό γραφειοκρατίας και κανόνων. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό πάρα πολύ. Αλλιώς μπορώ να συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε η κυρία Σεν του Τσέντεου Τσέσου και σας ευχαριστώ και πάλι για αυτή την ανοιχτή συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μπέγγελ. Τον λόγο λοιπόν τον επιστρέφω στην ευρωπαϊκή πλευρά και σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε να δώσετε τον λόγο στον επόμενο μιλητή. Ε, thank you very much. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ο μιλητής μας θα είναι ο σκιώδης ηγητής των φιλελευθέρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Κριστιαν Μπουζόη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που τελικά μας δίνεται η ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων με συναδέλφους από τον Bundestag για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα και μια και η συνεργασία μας είναι απαραίτητη για να βελτιώσουμε την ποιότητα και την εφαρμογή της νομοθεσίας μας. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο εξυγχρονισμός του συστήματος για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων είναι ε, επιτακτική ανάγκη προκειμένου να ενισχύσουμε την κινητικότητα των επαγγελματιών. έχουμε πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις από τη Γερμανία να ενισχύσουμε το σύστημα των δηλώσεων, να το πλουστεύσουμε για να ε, βελτιώσουμε τη μερική διπλο, ε, πρόσβαση. Σε ό,τι αφορά τους ε, συνοδούς, τους ξεναγούς, είναι σημαντικό να μην τους επιβάλλουμε το σύστημα δηλώσεων, γιατί δεν υπάρχει επαφή με τοπικούς καταναλωτές και άρα δεν διακυβεύεται η προστασία των καταναλωτών. Η επαγγελματική ταυτότητα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο για την προσωρινή κινητικότητα και θα μπορούσε ακόμη και να αντικαταστήσει στο μέλλον το σύστημα των δηλώσεων. Φυσικά χρειαζόμαστε ε, μελέτη επιπτώσεων αυτών των επαγγελματικών ταυτοτήτων και πάνω απ' όλα θα πρέπει να είναι προαιρετικές. Να εξετάσουμε και το θέμα της ε, κινητικότητας από ένα κράτος που δεν ρυθμίζει αυτό το θέμα σε ένα κράτος που το ρυθμίζει. Ε, η διετής επαγγελματική εμπειρία, είναι υπερβολικά επαχθή όρο. Σωστά η Γερμανία υποδεικνύει ότι οι επαγγελματίε που μόλι αποφύτησαν, οι πτυχιούχοι δεν μπορούν να αποδείξουν διαιτή επαγγελματική πείρα γιατί δεν μπορούν να τη συγκεντρώσουν. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε λύσει για τέτοιου περιπτώσει. περιπτώσεις. Και τέλο, το σύστημα για την αυτόματη αναγνώριση λειτουργεί ικανοποιητικά κατά τη γνώμη μου. Αλλά τα ελάχιστα οι ελάχιστε προποθέσει άσκηση ε, χρήζουν ενημέρωση και εξυγχρονισμού και μάλιστα τακτικά. Συμφωνώ με μια προσέγγιση που θα επικεντρώνεται στις δεξιότητες. Τα ελάχιστα, οι ελάχιστες προδιαγραφές άσκησης θα πρέπει να προσδιοριστούν όχι με βάση τη, μόνο τη διάρκεια της άσκησης, αλλά και τις γνώσεις, ώστε να προβλέπεται καλύτερη συγκρισιμότητα και να διευκολύνεται η διαδικασία αναγνώρισης. Γενικά θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να γίνουν και περαιτέρω βήματα για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο σύστημα και όταν το πετύχουμε αυτό θα είναι πολύ πιο εύκολο να σημειώσουμε και πρόοδο υπέρ της απλούστευσης για να εξυπηρετήσουμε και τους επαγγελματίες αλλά και τους καταναλωτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπουζόη. Θα ξαναδώσω το λόγο στον πρόεδρο από το Βερολίνο. Ευχαριστώ και θα δώσω τον λόγο αμέσως την κυρία Άτκενς Αλπέτς που είναι η εκπρόσωπος των αριστερών για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα συνάδελφοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την διεθνή συνεργασία και χαιρετίζω οπωσδήποτε την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας, αλλά μπροστά μας έχουμε κάποιες προκλήσεις. Ξέρετε πως ε, δεν παίζει σε πολλές ε, χώρες σημαντικό ρόλο η κουλτούρα υποδοχής και αναγνώρισης, αλλά και το πώς θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε τα γλωσσικά προσόντα των ανθρώπων που ε, θα πάνε σε άλλη χώρα να εργαστούν. Έτσι λοιπόν, για να είναι απλό και διαφανές το σύστημα αυτό της αμοιβαίας αναγνώρισης, θα πρέπει να δούμε ποιες δυνατότητες υπάρχουν για να μπορέσουν οι σχεδόν χίλιες αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας να περιοριστούν σε λιγότερες για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο συνοπτική διαδικασία. Επίσης, εάν αναγνωριστούν μόνο μερικά προσόντα, θα εξαρτάται μετά το εάν είναι δυνατόν η άσκηση του, να γίνει η άσκηση του επαγγέλματος από το εάν θα υπάρξει κάποια περαιτέρω εκπαίδευση. Αυτό ισχύει βεβαίω και για αυτού οι οποίοι είναι στην ίδια του χώρα και για αυτού οι οποίοι πάνε σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης. Επίση, οι επαγγελματικές αυτές ταυτότητες θα μπορούσαν να δείχνουν το μέλλον εάν είναι υποχρεωτική η αναγνώριση για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει πως θα έχουμε ελάχιστες υποχρεώσεις εκπαίδευσης για διάφορα κράτη-μέλη που θα πρέπει να αλλάζουν συνεχώς για να υπάρξει μία εγγύηση της ποιότητας. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μία αυτόματη αναγνώριση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη συντομία σας και δίνω τον λόγο ξανά στις Βρυξέλλες. Uh, thank you, Ευχαριστώ. Και ο τελευταίος μας σκιώδης ηγητής, η κυρία Χάιντι Ρούλε, που εκπροσωπεί τους Πρασίνους. κυρία Ρούλε έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Δυστυχώς βεβαίω εδώ πέρα θα έπρεπε να μιλήσει η συνάδελφός μου από τη Δανία, αλλά βρίσκεται σήμερα στην Κρακοβία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Γερμανούς συναδέλφους. Νομίζω πολλά από αυτά τα οποία είπαν σήμερα θα μπορέσουν να συνεισφέρουν στο έργο μας. Ειδικά όσον αφορά την ε, διάρκεια της ε, εκπαίδευσης ε, στον ανώτατο τομέα, γιατί δεν θα πρέπει βεβαίως να δώσουμε την εντύπωση πως οι άνθρωποι οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν λιγότερο θα πρέπει να έχουν κάποιο μειονέκτημα μετά στην αγορά εργασίας. Βλέπουμε λοιπόν πως οι παρατηρήσεις σας εδώ πέρα θα βρουν ε, φοροέδαφος, αλλά πρέπει να πούμε πως σημαντική είναι η συνεργασία μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί βεβαίως η εφαρμογή της οδηγίας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, έχει διαρκέσει πάρα πολύ και δεν ήταν και ολοκληρωμένη. Γι' αυτό είναι σημαντικό να δούμε ποιες είναι οι εμπειρίες που είχαμε για να αποφευχθούν στο μέλλον. Εάν δούμε ξανά τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή μιλάμε εδώ πέρα για τις προσφυγές ανθρώπων που αισθάνονται πως έχουν αδικηθεί, όπως παραδείγματος χάρη όταν κάποιοι πάνε στο Solvit, να το απλοποιήσουμε, να γίνει η διαδικασία λιγότερο γραφειοκρατική, αλλά βεβαίως πάντα με τη διασφάλιση της ποιότητας. Και έχει εδώ πέρα, νομίζω, μεγάλη σημασία το, η επαγγελματική αυτή ταυτότητα. Και βεβαίως χρειάζονται και κάποιες μελέτες εφαρμογής, αλλά νομίζω αυτή η επαγγελματική ταυτότητα ως ηλεκτρονική ταυτότητα έχει να προσφέρει πάρα πολλά στην επιτάχυνση και απλοποίηση της διαδικασίας. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστούμε κύριε Ρουλέ και ευχαριστούμε που τηρήσατε και το χρόνο αγόρευσης. Ξαναδίνω το λόγο στον πρόεδρο Χίνσκινγκ από το Βερολίνο. Θα περάσω στον κύριο Μεχμέτ Κίλιτς των Πρασίνων για της Πράσινης Ομάδας στην ε, Ομοσπονδιακή Βουλή. Έχετε το λόγο. Είστε αισιόδοξο κύριε Πρόεδρε ότι θα προλάβω, αλλά θα προσπαθήσω. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ την Κομισιόν για την αξιολόγηση της λειτουργίας και της εφαρμογής οδηγίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσώπων. Για ε, εμάς πέντε πράγματα έχουν σημασία. Πρώτα απ' όλα αποφυγή της γραφειοκρατίας. Υποστηρίζω βεβαίως το ότι θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των ε, επαγγελμάτων που ρυθμίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της αυτόματης αναγνώρισης. Δεύτερον, δεσμευτικότητα. Πράγματι, είμαστε υπέρ αυτού του εθελοντικού της εθελοντικής επαγγελματικής ταυτότητας, αλλά νομίζουμε πως θα πρέπει να υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες να ζητήσουν αυτό το χαρτί ή όχι. Και βεβαίως ε, σημασία μετά θα έχει να μπορούν να βασιστούν σε αυτό και να αποδείξουν και να αναγνωριστεί από τα άλλα κρατημέλη. Κατόπιν να έχουμε μια στοχευμένη δράση. Δεν θα πρέπει να χαθούμε στις λεπτομέρειες όταν μιλάμε για τις διάφορες φάσεις της εκπαίδευσης. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να εξετάσουμε το αν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές και πώς μπορούν αυτές να εξισωθούν. Τέταρτον, διαφάνεια. Ειδικά όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα και τα μέτρα εξίσωση, χρειαζόμαστε κριτήρια τα οποία θα είναι σαφή και κατανοητά από όλους πέμπτον και τελευταίο συνοχή. Εδώ πέρα θα ήθελα να τονίσω πως για μας έχει μεγάλη σημασία τα κράτη-μέλη να φροντίσουν και για την διευκόλυνση της αναγνώρισης ε, επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε τρίτες χώρες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Το ήξερα πως θα είστε σύντομος και θα μπαίνατε στην ουσία του ζητήματος. Σας ευχαριστώ κύριε Κίλιτς. Δίνω τον λόγο πάλι στην ευρωπαϊκή πλευρά σε σας κύριε Χάρμπορ. Ε, well, thank you, οι εισηγητές μας, συνεισηγητές μας από την αριστερά και την δημοκρατία και ελευθερία δεν είναι εδώ. Έχουμε τη διαδικασία Catch the Eye. Έχω τρεις θέσεις για ενός λεπτού ομιλίες. Έχουν ζητήσει το λόγο η κυρία Γκέπχαρντ, η Ριγκογέν και άλλη μία συνάδελφος. Μετά θα σας δώσω το λόγο Πρόεδρε και για τρεις παρεμβάσεις από δική σας πλευράς και μετά θα πρέπει να κλείσουμε γιατί έχουμε αρχίσει να καθυστερούμε. Δεν νομίζω ότι θα μας κλείσουν ακριβώς τις τέσσερις, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ζητήσω από την κυρία Ιρυμπογέν να ξεκινήσει. Παρακαλώ όμως σεβαστείτε το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας. Γεια σας, σας καλωσορίζω όλους. Σα χαιρετίζω όλους, όλους εγκαρδίως, ιδιαίτερα του συναδέλφου των Bundestag. Εμείς θα συμφωνήσουμε λέγοντας ότι η κινητικότητα των επαγγελματιών δεν είναι μόνο κάτι το οποίο προέρχεται από τις συνθήκες, αλλά είναι και κλειδί για την οικονομική ανάκαμψη και την οικονομική αηφορία. Οι τροποποιήσεις στην αγορά εργασίας είναι πολύ πιο γρήγορες από τις νομοθετικές μας ρυθμίσεις, γι' αυτό είναι απαραίτητο να προσπαθήσουμε να επικαιροποιήσουμε το σύστημα απόκτησης επαγγελματικών ικανοτήτων και να το προσαρμόσουμε στην πραγματικότητα της αγοράς εργασίας και στη ζήτηση. Όσοι πήραν το λόγο πριν από μένα λέγουν και συμφωνώ μαζί τους ότι θα πρέπει να στοχεύσουμε σε υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας, απλούστευσης των κανόνων και διευκόλυνσης της αμοιβαίας αναγνώρισης. Θα πρέπει να δούμε και ποια είναι τα αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία θα ληφθούν για να αντιμετωπιστούν τα υπάρχοντα προβλήματα και για να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται για τους επαγγελματίες. Πρέπει να εναρμονίσουμε τα κριτήρια τα οποία ισχύουν ιδιαίτερα στον τομέα τον γλωσσικό η Ευρώπη νομίζω ανήκει σε όλους, η ευθύνη για την Ευρώπη ανήκει σε όλους. Η Ευρώπη θα πρέπει τους επαγγελματίες και τους καταναλωτές να τους βάλει στο κέντρο, στην καρδιά της εσωτερικής αγοράς. Έτσι θα βγούμε από την κρίση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ριγκοϊένα. Η κυρία Βάιλερ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Χίντσκεν και συνάδελφοι, πρώην συνάδελφοι από την Ομοσπονδιακή Βουλή. Θα περιοριστώ σε τρία πράγματα, αλλά πρώτα απ' όλα να πω πως ακόμα και αν εμείς είμαστε εδώ πέρα Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς θα καταλάβατε πως για τους περισσότερους από εμάς το σημαντικότερο είναι το δικαίωμα των πολιτών να ασκήσουν ένα επάγγελμα ή να αναζητήσουν εκπαίδευση σε μια άλλη χώρα. Γιατί βεβαίως αυτό είναι σημαντικό για τους πολίτες. Υπάρχει και η αναγκαιότητα για την εσωτερική αγορά, αλλά πρώτα απ' όλα το θεωρούμε ένα δικαίωμα των πολιτών, να εργαστούν δηλαδή εκεί όπου θέλουν. Δεύτερον, σημαντικό είναι αυτό το οποίο είπε η κυρία Ρούλε, οι κυβερνήσεις ε, έχουν χτίσει πολύ περισσότερα τείχη από, όσα, ε, από όσο γνωρίζουν και από όσο γνωρίζουν οι βουλευτές ε, στα κράτη-μέλη, χωρίς να σημαίνει πως η Γερμανία είναι πρώτη. Και άλλα κράτη-μέλη το έχουν κάνει, αλλά πρέπει να μην ε, διαρκέσει αυτή η μεταρρύθμιση πολλά, πολύ χρόνια περισσότερα από όσο θα πρέπει. Και βεβαίως θα πρέπει να φροντίσουμε τα δικαιώματα και οι ιδιαιτερότητες ε, των χειρονακτικών επαγγελμάτων που μαθαίνουν δίπλα στο μάστορα οι νέοι να ε, διατηρηθούν. Αυτό έχει λειτουργήσει επιτυχώς σε Γερμανία, σε Λουξεμβούργο, σε άλλες χώρες και θα πρέπει να παραμείνει στην διαδικασία αυτή τη διαπραγματευτική και να μην διαλυθεί ξανά. Η κυρία Γκέπχαρντ, ηγέτη των σοσιαλδημοκρατών στη χώρα μας, στην ε, επιτροπή μα. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι στη Γερμανική Βουλή να επαναλάβω μια παρατήρηση ενός συναδέλφου. Πράγματι δεν θα πρέπει να μπει από την πίσω πόρτα ξανά η αρχή της χώρας προέλευσης. Ε, θέλουμε, θα το προσέξουμε αυτό γιατί οπωσδήποτε δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε. Πρέπει να φροντίσουμε τις δυνατότητες κινητικότητας που έχουμε να τις διαμορφώσουμε όσο δυνατόν πιο απλές. Και βεβαίως ε, εδώ πέρα το ζήτημα της επαγγελματικής ε, ταυτότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσο. Και βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις ε, αυτό ισχύει για τους αρχιτέκτονες, μηχανικούς, αλλά και για τα επαγγέλματα της υγείας, όλα αυτά που έχουν δηλαδή μεγάλη κινητικότητα, να τους δώσουμε την δυνατότητα έτσι ώστε να γίνει πιο απλούστερη η διαδικασία αυτή και να μπορούν γρήγορα να έχουν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Αυτό είναι το θέμα. Και βεβαίως ε, το έχουμε σκεφτεί αυτό σε μια εθελοντική βάση. Δεν μπορούμε να εξαναγκάσουμε κανέναν να έχει μια τέτοια ευρωπαϊκή ταυτότητα. Ίσως σε κάνα δύο αιώνες, ε, εν πάση περιπτώσει, να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά όπως είπα δεν θέλουμε να το κάνουμε υποχρεωτικό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ του τρει συναδέλφου για τη συντομία του, Θα δώσω τώρα το λόγο στον συμπρόεδρό μου στο Βερολίνο για να ακούσουμε και τις ομιλίες της δικής του πλευράς εφόσον το επιθυμών. Και μετά θα ακούσουμε μια σύντομη δήλωση του εισηγητή μας από τη μία και της Επιτροπής από την άλλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω τον λόγο αμέσως σε τρεις συναδέλφους, πρώτα απ' όλα στον κύριο Κάμπ, μετά στον κύριο Μπάρτλ και μετά στην κυρία και ελπίζω να έχουμε μετά χρόνο για να ακούσουμε και άλλες παρεμβάσεις καθώς ακόμα δεν έχει πάει τέσσερις. Κύριε Κάμπ, έχετε τον λόγο. Ο κύριος Κάμπ είναι μέλος του FDP των Φιλελευθέρων. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη. Να πω λίγα λόγια για το ευρωπαϊκό και το γερμανικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων. Εμείς εκτιμούμε την οδηγία αυτή που αποτελεί μέσο διεθνούς συνεργασία και βεβαίως υπάρχει μια συγκρισιμότητα όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα. Για εμάς λοιπόν είναι σημαντικό η ε, οδηγεί αυτή και το εθνικό πλαίσιο αναγνώριση προσόντων να γίνουν πιο λογικά. Θέλουμε βεβαίως, όπως είπαμε, μια ισοτιμία και μια διαφάνεια σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα πρέπει βεβαίως να διατηρήσουμε την υψηλή ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Γερμανία και να μπορέσει να μεταφερθεί με διάφανο τρόπο και στην Ευρώπη. Οι επαγγελματίε βεβαίω με τι ικανότητέ του είναι η κινητήριο δύναμη τη γερμανική οικονομία, Με αυτού βγήκαμε από την κρίση και βεβαίω ε, δίνουμε μεγάλο βάρο στο γερμανικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων και στην δυνατότητα λειτουργία του και στην Ολομέλεια τι ερχόμενε ημέρε, Οι Υπουργοί Παιδείας ε, των κρατηδίων θα ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Οπότε παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά το ζήτημα αυτό, το γερμανικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για να υπάρχει ε, δυναμική και κινητικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε, ο κύριος Μπάρτελ κατόπιν. Ένα λεπτό έχετε. Σας ευχαριστώ για την ε, συζήτηση αυτή. Να αναφερθώ σε κάτι που είπε ο Σον, γιατί δεν αναφέραμε κάτι για το κατόφλι της προϋποθέσεις της κοινή πλατφόρμας, γιατί νομίζω πως πρέπει να πούμε πως δεν θα πρέπει με ένα νέο κατόφλι να οδηγηθούμε στο ότι η μειοψηφία των κρατών μελών θα μπορέσει να μειώσει, αν θέλετε, το επίπεδο. Δεύτερο, είναι το ζήτημα της συγκρισιμότητας του χρόνου εκπαίδευσης. Εδώ πέρα έχουμε διαφορετικά μέτρα στην Ευρώπη, είτε είναι χρόνε, ώρες, έτη, τρίμηνα, εξάμηνα κτλ. για τον, χώρο, τον χρόνο με εκπαίδευση. Και τέλος η διαφάνεια και η αξιολόγηση προϋποθέτουν πως θα έχουμε μια διαδιακασία η οποία θα είναι διαρκής όσον αφορά αυτή την αξιολόγηση και θα εγγυάται έτσι πως ε, τα νέα κρατημέλη θα δηλώνουν τις νέες εξελίξεις στην Ευρώπη έτσι ώστε κάποιος ο οποίος ξεκινάει τις σπουδές του να γνωρίζει το τι γίνεται και το τι δυνατότητες έχει να δραστηριοποιηθεί αλλού εάν υπάρχει μια αναγνώριση των προϊόντων των προσόντων του μεσχόλου σε άλλη χώρα. Η κυρία Σεν έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Σύντομα θέλω να συμπληρώσω δύο πράγματα ε, από τους συναδέλφους από την Επιτροπή Υγείας οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορούν να είναι εδώ παρόντες σε σχέση με αυτό το οποίο είπε και ο κύριος ε, Μπάρτλ, είναι σημαντικό πράγματι η ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης για την βασική εκπαίδευση των ιατρών να είναι, όπως είπαμε, έξι έτη και επίσης το θέμα των φαρμακοποιών είναι πάρα πολύ σημαντικό, το τόνισαν όλοι οι συνάδελφοι από τον τομέα της υγείας ε, για την αυτόματη αναγνώριση των πτυχίων των φαρμακοποιών Εμεί, όπω και σε άλλες χώρες, ε, ξέρετε, υπάρχουν κάποια μονοπόλια σε αυτόν τον ε, τομέα και βλέπουμε πάρα πολύ δύσκολες οποιοσδήποτε αλλάγέ. Σα ευχαριστούμε κυρία Σεν. Κύριε Χάρμπορ, κύριε συνάδελφε, προτείνω τώρα να περάσουμε στις τελικές μας παρατηρήσεις για να μην ξεπεράσουμε και το χρόνο μας. Οπότε δίνω τον λόγο ξανά σε εσά για να μπορέσετε να ε, δώσετε τον λόγο στους συναδέλφους. Well, thank you very much, Chairman. Yes. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Ναι, και εγώ φοβόμαι ότι δεν προλαβαίνουμε να δώσουμε το λόγο σε άλλους ομιλητές γιατί σχεδόν εξαντλήσαμε το χρόνο που είχαμε για τη συζήτηση αυτή. Οπότε θα ήθελα να να παρακαλέσω του επόμενου ομιλητέ να περιοριστούν στο τρίλεπτο, τετράλεπτο το πολύ. Δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργαν Τρίτσερ που είναι ο τματάρχης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρμόδιος για το δοσχέ αυτό τη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Περιμένω τι δικέ του παρατηρήσει και κατόπιν θα ξαναδώσω το λόγο στην εισηγήτριά μα, την κυρία Μακλάρκιν, για να ανακεφαλαιώσει τα κεντρικά σημεία τη συζήτηση. και μετά θα σα ξαναδώσω το λόγο κύριε Πρόεδρε από την Bundestag για να ολοκληρώσετε. Κύριε Τίτσερ. Ευχαριστώ κύριε και κύριοι και η Κομισιόν ε, χαιρετίζει αυτή τη συζήτηση ε, και στο Κοινοβούλιο και στην Γερμανική Βουλή. Εμείς έχουμε πει πως ε, υπάρχουν πολλά σημαντικά και ευαίσθητα ζητήματα. Θα ήθελα εγώ να περιοριστώ τώρα σε τρία από αυτά. Το πρώτο είναι η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας ευχαριστούμε για τις απόψεις σας που μας στηρίζουν. Το πρόβλημα είναι όπως ξέρετε το τι γίνεται με τα κράτη-μέλη της υποδοχής. Εάν κινούνται γρήγορα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά συχνά το κράτος μέλος ε, δεν τηρεί αυτά τα οποία αναφέρονται στην ε, οδηγία. Οπότε δεν θα πρέπει να, δεν θέλουμε εδώ πέρα να ξαναφέρουμε την αρχή της χώρας προέλευσης, να δώσουμε μια δυναμική στην όλη διαδικασία. επίση αναφέρθηκε η πολυπλοκότητα του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων. Να σας πω εδώ πέρα πως το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων είναι ένα μέσο του τομέα εκπαίδευσης μέσω μιας σύστασης του 2008. Εδώ πέρα όμως είμαστε στον τομέα της εσωτερικής αγοράς και δεν μπορούμε να πούμε απλά πως είναι κάτι το δεσμευτικό. Εδώ πέρα υπάρχουν πολλά ερωτήματα στην πράξη. Η Κομισιόν ε, έχει κάνει μια μελέτη την οποία θα υποβάλει τέλος Οκτωβρίου. Το τρίτο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι η μερική ή τμηματική αυτή πρόσβαση. Δεν μου προξενεί έκπληξη πως υπάρχουν επικριτικές φωνές, αλλά να αναφέρω κάποια παραδείγματα. Φανταστείτε παραδείγματο χάρη μια Γερμανίδα νηπιαγωγό η οποία πάει στην Ολλανδία ή κάποιος ο οποίος ε, είναι ας πούμε μηχανικός και πάει στην Ισπανία χωρίς την μερική αυτή πρόσβαση δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Όπως σας είπα, είναι πράγματι επίμαχο, θα καταθέσω μια νομοθετική πρόταση στο τέλος του έτους και να αναμένουμε την, ε, να συνεχιστεί η θετική συζήτηση που είχαμε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Well, thank you very much Mr. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που είστε τόσο ε, συνοπτικός. Και τώρα θα ξανακούσουμε ε, την εισηγητριά μας, την κυρία Μακλάρκιν, για την ανακεφαλαίωση. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν και από το Βερολίνο και εδώ από τις Βρυξέλλες στη συζήτηση. Χαίρομαι για τη δέσμευσή σας ε, και για ε, το πόσο εξοικειωμένος είστε με το θέμα αυτό. Και χαίρομαι για το πώς επένδυσε και η γερμανική πλευρά σε αυτό το θέμα και επενδύσαμε στο ρόλο των κρατών μελών για να γίνει αποτελεσματική η εφαρμογή αυτής της οδηγίας και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην αναγνώριση του συστήματος επαγγελματικών προσόντων. Συμφωνώ απόλυτα, χρειάζεται streamline να γίνει το σύστημα πιο φιλικό προς το χρήστη, όσο πιο απλό γίνεται, να αξιοποιήσουμε τα επαγγελματικά προσόντα, προσόντα και τις δεξιότητες και να υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτά και εξασφαλιστεί στους επαγγελματίες η δυνατότητα ελεύθερης διακίνησης επίσης αναγνωριστεί η διαδικασία της Μπολόνια και να γίνει ανταλλαγή των πληροφοριών για την εκπαίδευση και αναγνώριση των διαφόρων μαθημάτων. Και αυτό το στοιχείο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Πάντω είναι προτεραιότητα το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι προτεραιότητα και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μία από τι προτεραιότητε του Επιτρόπου Μπαρνιέ για να προχωρήσει η, εσωτερική αγορά. Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική ταυτότητα, ε, Συμφωνώ ε, η πρόταση να είναι ηλεκτρονική αυτή η επαγγελματική ταυτότητα και φυσικά προαιρετική. Αλλά περιμένουμε και τη μελέτη επιπτώσεων αυτή τη επαγγελματική ταυτότητα και να, γίνεται, να γίνει μετά από βάση ανάλυση κόστου-οφέλου. Πάντω, εκτιμώ ιδιαίτερω ε, τα σχόλια που ακούσαμε από το Βερολίνο. Ήταν πολύ χρήσιμα και σα ευχαριστούμε και για το χρόνο που αφιερώσατε στη συζήτηση. Σα ευχαριστούμε, κύριε Μακλάρκινγκ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μα, όλου και όλου του που ήρθαν, αλλά και όσου έλαβαν μέρο στη συζήτηση. Και ιδιαίτερα θερμά ευχαριστώ προ τον Γιώργαν Τίτσερ, γιατί παρακολουθεί εκ του και στο θέμα. Και θα ήθελα ιδιαίτερω να ευχαριστήσω και το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και του διερμηνεί που χρησιμοποιούν αυτή τη νέα τεχνολογία και το συναρπαστικό είναι ότι περνάει μέσα από το ίντερνετ. Ε, γίνεται η αναμετάδοση μέσω του ίντερνετ, με πολύ απλό δηλαδή και προσιτό τρόπο. Και ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε κι εσείς ποια ήταν η εμπειρία από αυτό, είναι τα χρήσιμα, γιατί θα ήθελαμε να επαναλάβουμε τέτοιες εμπειρίες και με τη δική σας Βουλή, αλλά και με άλλα κοινοβούλια και άλλες επιτροπές. Πάντως πραγματικά ήμασταν πρωτοπόροι στη δοκιμασία αυτού του τρόπου τις τεχνολογίες και νομίζω ότι και η Ειδική Επιτροπή χαίρεται για την πρωτοπορία αυτή και τη χρήση των νέων τεχνολογιών σε αυτή την επικοινωνία. Ευχαριστούμε θερμά τους εκπροσώπους του Bundestag και δίνω το λόγο στον ε, πρόεδρο από το Bundestag για τα τελικά σχόλια. Σας ευχαριστώ και εγώ κυρία Χάρμπορ ε, για το ότι μου δίνετε την δυνατότητα να παρέμβω. Να ευχαριστήσω και εγώ πράγματι τους διερμηνείς που εργάστηκαν εξαιρετικά και πράγματι απέδειξαν πως έχουν τα επαγγελματικά προσόντα τα οποία εκτιμούμε και εμείς στη Γερμανία όπως και οι Ευρωπαίοι γειτονές μας. Δεύτερη παρατήρηση, θεωρώ πως ακριβώς αυτή η συζήτηση ε, σε νέα πράγματα τα οποία νομίζω μπορούν να αποτελέσουν βάση των διαβουλεύσεων στις επιτροπές μας. Τρίτον, στο μέλλον ακριβώς αυτό το οποίο ε, γάγαμε εμείς εδώ πέρα ως ε, Επιτροπή Τεχνολογίας να δημιουργήσει σχολή και να το υιοθετήσουν και οι υπόλοιποι γιατί με αυτό τον τρόπο νομίζω μπορούμε να συζητήσουμε τα διάφορα προβλήματά μας και να συνεργαζόμαστε εντατικά. Και τέλος, αναφερθήκατε σε τρία σημεία. Πρώτον, την ευρωπαϊκή ε, ταυτότητα και την ε, πρόσβαση. Κοιτάξτε, πράγματι το ζήτημα λοιπόν είναι ακριβώς αυτά τα οποία αναφέρατε και είναι και ευρωπαϊκό και εθνικό και Γι' αυτό ισχύει αυτό το οποίο είπε η κυρία Μακλάρκιν, ότι δηλαδή επιθυμεί ακριβώ αυτή η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα να είναι απλή και μη γραφειοκρατική, έτσι ώστε οι συμπολίτε μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, είναι και ικανοποιημένοι από την Ευρώπη γιατί θα είναι λιγότερο γραφειοκρατική από όταν σου παρελθόν. Σας ευχαριστώ λοιπόν, καλή σας επιτυχία και αναμένουμε την επόμενη συνομιλία μας. Πολύ αυθόρμητο αυτό το χειροκρότημα από εμά. Σα αποχαιρετούμε λοιπόν προ το παρόν, γιατί έχουμε κάποιε ψηφοφορίε που θα πρέπει να γίνουν. Πάντω, σα ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Uh, um, Συνάδελφε, νομίζω ήταν πολύ επιτυχημένη και συναρπαστική αυτή η βιντεοδιάσκεψη και η ευκαιρία που είχαμε και σας ευχαριστώ θερμά όλους για τη συμμετοχή σας. Νομίζω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να επαναληφθεί αυτή η εμπειρία. Γιατί ήταν πραγματικά μια άριστη ανταλλαγή απόψεων. Και μπορούμε να οργανώσουμε αντίστοιχη και με άλλες εθνικές βουλές. Περνάμε στις ψηφοφορίες. Πρώτα απ' όλα όμως κάποια διαδικαστικά. Καταρχήν να, ε, να κηρύξω την έναρξη, την επίσημη έναρξη της συνεδρίασης, να εγκρίνουμε και την ημερήσια διάταξη που έχει μοιραστεί. Φαντάζομαι όλοι θα συμφωνείτε. Δεν ξέρω αν έχουμε πρακτικά προσέγγιση, μάλλον όχι. Έχουμε και αναμετάδοση μέσω ίντερνετ και είχαμε και το newsletter της περασμένης εβδομάδας. Όσοι δεν προλάβατε την περασμένη εβδομάδα μπορείτε να λάβετε το αντίγραφο εδώ. Και στους θεατές από το ίντερνετ μπορείτε να μπείτε στο mailbox της Επιτροπής μας και να λάβετε εκεί το newsletter. Έχουμε αντίγραφο και στα γραφεία μπορείτε να τα μοιράσετε στους επισκέπτες σας, φαντάζομαι όλοι. Θα περιμένετε διακάως αυτή την ευκαιρία. Ετοιμαστείτε τώρα για την ψηφοφορία της ε, έκθεσης Μακλάκιν. Αρχικά δεν είχε προγραμματιστεί η ψηφοφορία αμέσως μετά την βίντεο διάσκεψη. Αρχικά είχε προβλεφθεί πριν από τρεις εβδομάδες ε, όταν έγινε η διακοπή ρεύματος στο blackout. Αλλά θα ψηφίσουμε τώρα. κυρία Μακλάρκιν, αν έχει κάποια σχόλια πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. Μια και όλο το απόγευμα συζητήσαμε αυτό το θέμα αυτό και εκτεταμένα και τους προηγούμενους μήνες, θα είμαι λακωνική. Να ευχαριστήσω θερμά τους και ηγητές. Ήταν πραγματικά μεγάλη χαρά τη συνεργασία μου μαζί του. Λυπάμαι τελευταία στιγμή ζητήθηκε ψηφοφορία κατά τμήματα σε ορισμένε τροπολογίες, γιατί εγώ νομίζω ότι αντικατόπτριζε ο κατάλογος των ψηφοφοριών και η πλήρης ε, μελέτη επιπτώσεων. Ελπίζω πάντως ε, στι υπόλοιπε τροπολογίες να συγκεντρώσουμε συντριπτική πλειοψηφία ώστε πραγματικά να έχω μια σχετικά στεναρή έκθεση για να είναι και χειρό το μήνυμά μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια και για το άοκνο έργο σας για την έκθεση αυτή. Θα ψηφίσουμε λοιπόν, θα έλεγα να κάνουμε μια δοκιμή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Συμβιβαστική τροπολογία 1, άρχεται η ψηφοφορία. 31 κάρτες μόνο έχουν εισαχθεί στο μηχάνημα. 32. Έχετε όλοι τις κάρτες. 32. 32 τελικά. Τέλος ψηφοφορίας. 32 υπέρ. Ωραία. Και εγκρίνουμε τη συμβαστική τροπολογία 1. Τροπολογία 19 του κυρίου Γκρέχ. Ποιος είναι υπέρ κατά εγκρίνεται. Επιτροπή Απασχόλησης, τροπολογία 1, ποιος είναι υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Επιτροπή Απασχόλησης, τροπολογία 2, υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος. Εγκρίνεται 18 υπέρ 13 κατά. Τροπολογία 26 Επιτροπής Απασχόλησης. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Μερικοί καθυστερούν πολύ να πατήσουν τα κουμπιά. Κάποιος δεν πρόλαβε να ψηφίσει. 16 υπέρ 15 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21 της κυρίας Βερνιό. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20 πολλών συναδέλφων. Ποιος είναι υπέρ. Άρχεται ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την τροπολογία 20. Ως προσθήκης. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 29. Τέλος. Εγκρίνεται. Τέταρτη τροπολογία της Επιτροπής Απασχόλησης. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται με σαφή διαφορά. Συμβαστική τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ κατά εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 44. Ποιος είναι υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 36. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 45. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται και αυτή. τροπολογία της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Όχι, καταπίπτει δεν χρειαζόταν καν, γιατί εγκρίθηκε 45. Τροπολογία 46. Ποιο είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, με σαφή διαφορά. Τροπολογία 51. ποιο είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 52. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται με διαφορά. Συμβαστική τροπολογία 7. Ζητήθηκε ψηφοφορία κατά τμήματα από τους πράσινους. Ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα της συμβαστικής τροπολογίας 7. Ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται γι' αυτό. Περνάμε στην τροπολογία 50... Στην, μάλλον στη 14η τροπολογία της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Έμβη 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 56. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 58. Υπέρ. Ε, μάλλον ηλεκτρονική ψηφοφορία. άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 59. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 124 καταπίπτει. Τροπολογία 60 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 61. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 62. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την 62. Τέλος. Εγκρίνεται. 19 ψήφι υπέρ, 14 κατά. Συμβαστική τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 70. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Για το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 70. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τώρα της τροπολογίας 70. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά, παρόλο που είμαι σχεδόν σίγουρο ότι εγκρίνεται, άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 70. Τέλος, σαφώς εγκρίνεται 19 υπέρ, 4 κατά. Συμβαστική τροπολογία 9, ψηφοφορία κατά τμήματα, τρία τμήματα, τα έχετε στον κατάλογο ψηφοφορίας. Κύριε Πρόεδρε, μόλις έρχομαι από την Επιτροπή Οικονομικών και εκεί πέρα διαπίστωσε ο Πρόεδρος πως δεν μπορούν να υπάρξουν πλέον περισσότερο, περισσότερες συμβιβαστικές ε, τροπολογίες με χωριστές ψηφοφορίες. Συμφωνείτε κι εσείς με αυτό για να δούμε, γιατί αυτό κάναμε μέχρι τώρα. Well, I think I'm entirely... σε εσά στις πολιτικές ομάδες. εγώ θα πρότεινα να το συζητήσουν στην επόμενη συνεδρίαση Σύμβουλη των Ομάδων και αν θέλουν να συμφωνήσουν να αποφεύγουμε ψηφοφορίες κατά τμήματα συμβαστικές τροπολογίες, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Ας το ανακοινώσω στη γραμματεία. Επίσης, αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα ε, θα πρέπει να γίνονται εγκαίρως και να μην υποβάλλονται τελευταία στιγμή. Από ό,τι ξέρω αυτό συμφωνήθηκε με, το, με την εισηγήτρια και τους υπόλοιπους, οπότε θα το εφαρμόσουμε. Νομίζω πως οι εμβαστικές ε, τροπολογίες κατευθύνται πάρα πολύ αργά και πρέπει να έχουμε και χρόνο να, τα, να τις δούμε. Δεν μπορεί μία ομάδα να μην συμφωνεί με ένα τμήμα της ε, τροπολογίας. Εντάξει, σε αυτή την περίπτωση είναι φυσιολογικό να ζητάει χωριστή ψηφοφορία. Δεν θέλω να περιορίσουμε τα δικαιώματα των βουλευτών και δεν πρέπει ε, οπωσδήποτε να έχουμε πάρα πολύ συχνά αυτές τις ε, καταστάσεις και να γίνει καθεστώς. Αλλά δεν νομίζω πως υπάρχει λόγος να το συζητήσουν οι συντονιστές. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το δικαίωμά μας. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ζητήθηκαν ψηφοφορίες κατά τη μάτα γιατί μόνο την ε, Παρασκευή το απόγευμα, το βράδυ σχεδόν, λάβαμε τις συμβαστικές τροπολογίες και είχαμε ελάχιστο χρόνο για να τις μελετήσουμε. Ναι, αντιλαμβάνομαι την πίεση. Εγώ δεν έχω τήρηση να, να κάνω ότι μου πούν οι ομάδες. Και έστω και κάποιες μερικές μικρο... Ε, μικροδιορθώσεις τελευταίες στιγμής αν εξυπηρετούν τις ομάδες δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, ας ψηφίσουμε κατά τμήματα, αναφέροντας στον κατάλογο ψηφοφορίας. Πρώτο τμήμα της συμβαστικής τροπολογίας 9. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9 και πάλι δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ε, απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Και τρίτο τμήμα της συμβαστικής τροπολογίας 9. Κατά. Εγκρίνεται και αυτό. Οπότε περνάμε στην τροπολογία 81. Άρχεται η ψηφοφορία για την 81. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 84. Άρχεται η ψηφοφορία για την 84. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 86. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 87 και 23 της Επιτροπής Περιβάλλοντος Πανομοιότυπες. Άρχιδη ψηφοφορία για τις δύο τροπολογίες. Τέλος. Απορρίπτονται. Συμβαστική τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 94. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Εγκρίνεται. 95 και 24 της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Εγκρίνονται. Συμβαστική τροπολογία 12. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 100. Κατά εγκρίνεται. 103 ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13 και πάλι ψηφοφορία κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το τμήμα 1 της 13, ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται και αυτό. Τροπολογία 109. Άρχεται η ψηφοφορία για την 109. Τέλος. Απορρίπτεται. 16 υπέρ 17 κατά. Τροπολογία 110. Άρχεται η ψηφοφορία για την 110. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 111. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 112. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 113 ως προσθήκη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13 καλύπτεται. Τροπολογία 114. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 116 λέει ο πρόεδρος. Όχι, 115, συγγνώμη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 116. Ποιος είναι ή μάλλον ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για την 116. Τέλος. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 118. Άρχεται ψηφοφορία για την 118. Τέλος. Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. 17 υπέρ, 15 κατά. Τροπολογία 117 ως προσθήκη. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22 της Επιτροπής Απασχόλησης καταπίπτει. Τροπολογία 119. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 14. Και πάλι κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 14, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 123. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 126 καταπίπτει και η τροπολογία 9 της Επιτροπής Απασχόλησης το ίδιο. Συμβαστική τροπολογία 15. Κατά τμήματα, πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτή. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Εκατόν σαράντα τρία. Αρκετά μπροστά. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ της 143. Κατά. δεκτεί. 145. Ποιοι είναι υπέρ. Δεκτή. Περνάμε τώρα σε αιτιολογικές σκέψεις. 1, 2 και 3, Ταυτόσιμες. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτές. Περιβάλλον 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περιβάλλον 5. Ποιοι είναι υπέρ κατά, δεκτή. Περιβάλλον 6, ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτή. Περιβάλλον 8, υπέρ, κατά, δεκτή. 4, υπέρ, κατά, δεκτή. 5, υπέρ, κατά, δεκτή. 6, υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία για την 6. Τέλος. Έχουμε και το Σκοτ Σόπλινγκ να ψηφίζει, απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 8 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 9. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την 9. Τέλος. Δεκτή. 18 υπέρ 14 κατά. Τροπολογία 10 υπέρ κατά. Δεκτή. 11 υπέρ κατά. Δεκτή. 12 υπέρ κατά. Δεκτή. 13 υπέρ κατά. Δεκτή. 14 υπέρ κατά. Δεκτή. 15 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περιβάλλον. Αιτιολογική σκέψη α υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έχουμε το β. Μπορώ να τις ψηφίσουμε ομαδών παρακαλώ. Όχι λένε οι βουλευτές. Λοιπόν β. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Σ αγγλικό υπέρ. Κατά Απορρίπτεται. D αγγλικό υπέρ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το D της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ή e, της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. F της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. G της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. H της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Και I της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται και αυτή. Σας ευχαριστώ όλους. Τώρα θα κάνουμε την τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ξεκινάμε. Πέρα στις ψηφοφορίες. 32 υπέρ, μία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Μακλάκεν. Εξαιρετική δουλειά. Όπως κάναμε ήδη και στο παρελθόν, θα γίνει μια συζήτηση και στην Ολομέλεια όπως είχε γίνει στην έκθεση της κυρίας Ρούλε. Νομίζω ότι θα το συζητήσουν και θα αποφασίσουν οι πολιτικές ομάδες. Η επόμενη ψηφοφορία μας είναι η ψηφοφορία της εκθέσεως του κυρίου Τριανταφυλλίδη. Θέλετε το λόγο κύριε Τριανταφυλλίδη πριν ξεκινήσουμε. Ευχαριστήσω τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν υποβάλει πάρα πολλές τροπολογίες και εμπλούτησαν το κείμενο της έκθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους εκπροσώπους της Κομισιόν, τη Γραμματεία της Επιτροπής μας, το προσωπικό των πολιτικών ομάδων, τους βοηθούς των συναδέλφων βουλευτών, τους σκιώδης εισηγητές. Ήταν μια έκθεση η οποία ε, προκάλεσε πολλές ε, φιλοσοφικές σκέψεις και την υποβολή είναι 128 τόσων ε, τροπολογιών με τη συνεργασία όλων κατορθώσαμε να κάνουμε αρκετές ε, compromise amendments. Ελπίζω ότι και η τελική ψηφοφορία θα αντανακλά αυτήν τη συλλογικότητα και να γίνει μια έκθεση της Επιτροπής και όχι του Κυριάκου Τριανταφυλλίδη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τριανταφυλλίδη για το πνεύμα συνεργασία του. Να κάνω μια σύντομη παρατήρηση. Θα ήθελα να τεθεί σε ψηφοφορία ένα τμήμα τη τροπολογία μου 45 που συνυπέγραψα με τον συνάδελφο Σφάμπ. Πρέπει να γίνει αυτό γιατί αυτό το τμήμα της 45 δεν καλύπτεται από τη συμβιβαστική 3. Αν θέλετε λοιπόν θα πρέπει να θέσετε σε ψηφοφορία τις τελευταίες ουσιαστικά λέξεις της τροπολογίας 45 χωρίς να δημιουργούνται επιπλέον εμπόδια για τις, ή βάρη για τις ε, επιχειρήσεις. Συμφωνείτε κύριε Τριανταφυλλίδη. Συμφωνείτε όλοι. Καλώς λοιπόν. Να μου το θυμίσετε όταν φτάσουμε εκεί. Ξεκινάμε την ψηφοφορία λοιπόν. 35. Θα ήθελα να βοηθήσω να επιταχύνουμε τη διαδικασία οι WIPs των πολιτικών ομάδων των δύο μεγάλων. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ 35, κατά, δεκτή, 36, υπέρ, κατά απορρίτεται. All the other ones fall, Okay. Uh, amendment 38. 38 υπέρ κατά δεκτή. 37 σαν προσθήκη. Ποιοι είναι υπέρ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 40. Ψηφίζουμε την 40. Απορρίπτεται. 39. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Οικονομική 2. Προσθήκη ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Πηγαίνουμε στην 188 Ροσφόρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Οικονομική 19. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Οικονομική 20. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 45 με την συμπληρωματική διευκρίνηση που έκανε η κυρία Λεγκρίπ. Για την 45 ψηφίζουμε. 45 συμπληρωματική διατύπωση. Α, για μια στιγμή λέει ο πρόεδρος. Η κυρία Λεγκρίπ προτείνει Θέλετε άμα ξαναπείτε τι προτείνετε κυρία Λεγκρίπ για να είμαστε σίγουροι. Θέλετε να είναι προσθήκη στην συμβιβαστική 3. Οι τελευταίες λέξεις της τροπολογίας σας να είναι συμπλήρωμα προσθήκη ε, στην 3 συμβιβαστική. Λοιπόν, τμήμα της 45 ε, ε, λοιπόν ψηφίστηκε Γίνεται δεκτή η πρόταση της κυρίας Λεγκρίπ. Περνάμε τώρα στην 54. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτή. Οικονομική 3. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτή. Συμβιβαστική 4. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτή. Περνάμε στη συμβιβαστική 5. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτή. Ψηφίζουμε τώρα για την 62 και 63 ως προσθήκη. Ποιοι είναι υπέρ. Ή μάλλον ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 62 και 63 προσθήκη. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 41. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 65. Ποιοι είναι υπέρ ποιοι είναι κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 6. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε τώρα στην 71. Με μια προφορική τροπολογία. Βλέπετε το κείμενο στο τέλος του κειμένου. Υπογραμμισμένο. Λοιπόν, 71. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 73. Head. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. Απορρίπτεται. 19 κατά 14 υπέρ. Συμβιβαστική 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε τώρα στην 81. Υπέρ κατά δεκτή. 82 υπέρ κατά δεκτή. 83 υπέρ κατά δεκτή. Θέλετε να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 83. Τέλος. Λοιπόν, 17 υπέρ, 16 κατά δεκτή. Λοιπόν, συμβιβαστική 8, ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτή. Πηγαίνουμε τώρα στην συμβιβαστική 9, ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτή. Και στην 84, Ξεχωριστή ψηφοφορία. Έχει ζητηθεί από το ΕΛΚ. Θέτουμε σε ψηφοφορία τώρα το πρώτο τμήμα της 84. Το πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. 21 υπέρ 12 κατά δεκτή. 84 δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτό. 94. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 72. Ποιοι είναι υπέρ. Ή μάλλον ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 72. Τέλος. Απορρίπτεται. 95. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 97. Άρχεται η ψηφοφορία για την 97. Απορρίπτεται. 96. Προσθήκη. Καταπίπτει μάλλον αυτή. 98. Γκρέτς. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 99 υπέρ της 99 κατά δεκτή 100 υπέρ κατά απορρίπτεται 102 Άρχεται η ψηφοφορία για την 102. Πέρας της Απορρίπτεται. 101 οικονομική 22. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτές. Οικονομική 23 προσθήκη ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Οικονομική 24 προσθήκη ποιοι είναι υπέρ. Δεκτή. Πηγαίνουμε συμβιβαστική 10 Ξεχωριστή ψηφοφορία, όπως έχει ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και την ομάδα των συντηρητικών. Λοιπόν, πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτή. Συμβιβαστική τροπολογία δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονική ψήφος. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά το δεύτερο τμήμα της 10. Περνάμε λοιπόν τώρα στην οικονομική 12. Προσθήκη. Οικονομική 12. Ποιοι είναι υπέρ. Ή μάλλον ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την οικονομική 12. Τέλος. Δεκτή. Περνάμε στην τροπολογία 109. Λεγκρίπ και Σβάμπ. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. 19 υπέρ 13 κατά. Οι υπόλοιπες καταπίπτουν. Γιατί αυτή διέγραφε πολλές. Πηγαίνουμε στην 118 τώρα. Head. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 118. Τέλος. Απορρίπτεται. Περνάμε συμβιβαστική 11. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 124. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 125 και 126 Α, έχουν καταπέσει αυτές λόγω της συμβιβαστική. Περνάμε λοιπόν στην 133, 134 και 135 που διαγράφουν άλλες παραγράφους. Λοιπόν, ψηφίζουμε τις τρεις από κοινού. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος, δεκτές. Όλες οι υπόλοιπες τροπολογίες της 17 καταπίπτουν και περνάμε τώρα στην 140. Πάξας. 140. Ποιοι είναι υπέρ ή μάλλον ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. Απορρίπτεται. 170. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Έχουμε την τροπολογία 141, 142, 143. Ψηφίζουμε από κοινού. Τέλος. Οι 144 καταπίπτει γίνονται δεκτές. Πηγαίνουμε τώρα στην 147. Είναι υπέρ, κατά. Δεκτή. 148. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 148. Τέλος. Απορρίπτεται η 148. Οικονομική 6. είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Οικονομική 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Όχι, όχι, όχι. Η οικονομική 9. Άρχεται η ψηφοφορία για την 9. Τέλος. Δεκτή. Οικονομική 10. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά την 10 της Οικονομικής Επιτροπής. Τέλος. Οικονομική 16. Τέλος. Δεκτή με μία ψήφο. Διαφορά. 149. Ροσφό. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 150. Ποιοι είναι υπέρ. Ή μάλλον ηλεκτρονική ψήφος για την 150. Αρχίζουμε. Τέλος. Δεκτή νομίζω ότι οι υπόλοιπε καταπίπτουν. Πηγαίνουμε λοιπόν στην 153 του κυρίου Ροσφόρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 13. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Πηγαίνουμε τώρα στην 157 της κυρίας Head. Ποιοι είναι υπέρ. Ή μάλλον ηλεκτρονική ψήφος για την 157. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική 12. Ποιοι είναι υπέρ. Όχι. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 12 πάλι. Διορθώνει ο πρόεδρος. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική 14. Ο Κυριάκος έχει το λόγο να διευκρινίσω, λέει ο κ. Τριανταφυλλίδης, ότι μετά τη συμβιβαστική ζητήθηκε την τελευταία στιγμή και χωρισμένη ψηφοφορία. Αυτό δεν μου έδωσε τη δυνατότητα να διαπραγματευτώ μια άλλη συμβιβαστική. Δεν είχαμε χρόνο να το κάνουμε. Και αυτή και χωρισμένη ψηφοφορία, εφόσον προχωρήσει, αφαιρεί μια πολύ βασική έννοια, την οποία θα ήθελα εγώ να αφήσω. Αλλά το αναφέρω αυτό όπως είπα οι προτάσεις αυτές που έρχονται την τελευταία στιγμή είναι προβληματικές. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εμένει στη σύστασή του, εκτός αν θέλετε να αλλάξετε κάτι την τελευταία στιγμή, στην Ολομέλεια ίσως. Αποσύρετε δηλαδή το έτοιμά σας για και χωρισμένη ψηφοφορία. Τι θέλετε να κάνετε ακριβώς, ρωτάει το ΕΛΚ. Όχι, παραμένει το αίτημα του ΕΛΚ, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται στις ψηφοφορίες ο τόπος που προτείνεται. Πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ τη συμβιβαστική 14 πρώτο τμήμα, δεκτή. Το δεύτερο τμήμα, ηλεκτρονική ψήφος για το δεύτερο τμήμα. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 167 ως προσθήκη του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ ή μάλλον ηλεκτρονικά καλύτερα για την 167 άρχεται ψηφοφορία. Η 167 ως προσθήκη στη συμβαστική. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με εμφανή διαφορά. Τροπολογία 166. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 168. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 169. Ως προσθήκη. Ποιος είναι υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία για την 169. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 171 του κυρίου Ρέπο. Ποιος είναι? Ή μάλλον ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία για την 171. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 173. 173. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 172. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. 174. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται και αυτή. 13. Τροπολογία της ΕΚΟΝ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. 175. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 176 καταπίπτει. 177. Ποιος είναι υπέρ. 177. Άρχεται η ψηφοφορία για την 177. Ποιος είναι υπέρ σε 177 κατά εγκρίνεται. Η 176 κατα... κατέπεσε. 178 του κυρίου Μότι. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται με διαφορά. Τροπολογία 179. Ποιος είναι υπέρ. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 179 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 180. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 181. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται και αυτή. 182. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την 182. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται με μία ψηφοδιαφορά. 18 της ΕΚΟΝ ως προσθήκη στην τροπολογία ΡΕΠΟ. Τροπολογία 18 της Οικονομικής Επιτροπής. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Πέρασε και η 182 και η 18 της Οικονομικής Επιτροπής. Τροπολογία 26 της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος. Εγκρίνεται τροπολογία 27 της ΕΚΟΝ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος εγκρίνεται και αυτή. 28 της Οικονομικής Επιτροπής ως προσθήκη άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 183. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος απορρίπτεται. 184, ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 186, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 185, ποιος είναι άκτη ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος. Εγκρίνεται με μία ψηφοδιαφορά. 187 κατά πίπτη, αν δεν κάνω λάθος, λέει ο Πρόεδρος. Όχι, όχι, θα την ψηφίσουμε ως προσθήκη στην 185. Τροπολογία Head, 187. Ποιος είναι υπέρ, ως προσθήκη. Υπέρ και πάλι, λέει ο Πρόεδρος, κατά αποχές Μάλλον ηλεκτρονική ψηφοφορία καλύτερα γιατί δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε την 187 προσθήκη της κυρίας Χέντ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις τώρα. Τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Δεκατρία. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Δεκατέσσερα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 4. Τροπολογία της ΕΚΟΝ. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. ΕΚΟΝ 5 υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 16. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 16. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά τμήματα. Το σύνολο του κειμένου πλην των λέξεων δικαιώματα, rights. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και το δεύτερο τμήμα, ο, τον όρο δικαιώματα δηλαδή, άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα, για τη λέξη δικαιώματα. Τέλος ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Τροπολογή 25, ποιος είναι υπέρ, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 25. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 της ΕΚΟΝ ως προσθήκη. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Εγκρίνεται με διαφορά. Τροπολογία 26. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 27. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Εγκρίνεται και αυτή. 28 με 30 ταυτόσημες ως προσθήκες. Άρχεται η ψηφοφορία για 28-29-30. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 31 για την τελική σκέψη. Α, ποιος είναι υπέρ. Άρχεται ψηφοφορία μάλλον ηλεκτρονικά. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32, όποιο είναι υπέρ, κατά. Εγκρίνεται 34 υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για τον 34. Τέλος. Με μία διαφορά εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, εγκρίνεται και αυτή. 7 ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 7 άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τελική ψηφοφορία για το σύνολο της έκθεσης. ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία για την έκθεση όπως έχει τροποποιηθεί. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ, καμία ψήφο κατά και 10 αποχές. Σας ευχαριστούμε κύριε Τριανταφυλλίδη. Φαντάζομαι θα έχουμε και άλλη δουλειά πριν την Ολομέλεια. Πολύ σημαντική όμως έκθεση. Κύριε Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ, Μάλκομ η ομάδα μου με παρακάλεσε στο τέλος της ε, ψηφοφορίας να αιτιολογήσω το γιατί ε, απήχαμε. Είναι καλή η έκθεση βεβαίως και θέλουμε να συμφωνήσουμε γιατί υπάρχει πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ μέσα αλλά λείπουν κάποια ουσιαστικά πράγματα τα οποία χάσαμε στην ψηφοφορία. Το ένα ήταν ε, οτιδήποτε είχε σχέση με την προστασία των παιδιών στην διαφήμιση. Και αυτό διαγράφηκε μέσω της τάσης των συντηρητικών και φιλελευθέρων. Αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Δεύτερον, διαγράφηκε οτιδήποτε είχε σχέση με τα κοινωνικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και ούτε με αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι για την Ολομέλεια. Γιατί δεν θέλουμε να έχουμε μισά πράγματα στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Well, thank you very much. Uh, well, I hope that we can. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να γίνει κάποια συζήτηση για να έχουμε και καλή πλειοψηφία. Έχετε δίκιο. Κύριε Σφάμπ. Και κύριε Πρόεδρε θα είμαι σύντομο. Και εμείς το ΕΛΚ υπερψήφισε στο τέλος παρά το ότι δεν πήγαν όλα όπως θέλαμε, αλλά ελπίζω να λυθούν τα ανοιχτά ζητήματα. Το ζήτημα δικαιωμάτων των εργαζομένων και άλλα σημαντικά ζητήματα δεν νομίζω όμως οπωσδήποτε πως πρέπει να λυθούν στη στρατηγική των καταναλωτών. Γι' αυτό επικεντρωθήκαμε στα βασικά και σε αυτά που ε, ανήκουν εδώ πέρα. Αλλά όπως ε, είπα νομίζω πως μπορούμε στη συζήτηση να βρούμε κάποιες ε, συμβαστικές λύσεις. Ευχαριστώ. Well, I rely all... Είμαι σίγουρος πως ε, με συνένεση και συνεργασία θα έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα και είναι σημαντικό για να θέσουμε κάποια ορόσημα για το στρατηγικό έργο της ε, Κομισιόν. Αλλιώς η Κομισιόν δεν θα λάβει υπόψη τα όσα λέμε. Λοιπόν, τώρα περνάμε στην έκθεση της κυρίας Κοράτσα Μπίλτ. Πρόκειται για γνωμοδότηση για την τροφή Περιβάλλοντος για το πώς θα αποφευθεί η σπατάλη τροφίμων. Θα δώσω λόγο στην εισηγήτρια να μας πει για τη ψηφοφορία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν ευχαρίστησή μου να εργαστώ πάνω σε αυτή την έκθεση και ευχαριστώ τους συναδέλφους για την στήριξη. Οι τροπολογίες ενίσχυσαν ε, την έκθεση για να μπορέσουμε περισσότερο, όχι ως νομοθέτες, αλλά ως διαμορφωτές της γνώμης. Για πρώτη φορά, εδώ πέρα δίνουμε τη δύναμη στους καταναλωτές και δεν τους διατάζουμε. Λέμε στους καταναλωτές, στο λαό της Ευρώπης, πώς μπορεί να κάνει τη διαφορά στην κουζίνα του, στο πώς ψωνίζει, στο πώς τρώει, στο εστιατόριο, τη θερμοκρασία του ψυγείου του. Μπορεί να κάνει την διαφορά με το να προωθήσει την υπεύθυνη και ε, φόρο κατανάλωση. Νομίζω λοιπόν πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ε, σημαντική αυτή η ηθική πτυχή σε μια εποχή όπου έχουμε προκλήσει οικονομικές, περιβαλλοντικές και ασφάλειας τροφίμων. Επίσης, ζητάμε και από τα εμπλεκόμενα μέλη να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη. Πολλά συμβαίνουν και βεβαίως πρέπει να ανταλλάξουμε ευέλτιστες πρακτικές ε, να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε και τα παιδιά σχολείο για τον πλαστικό πολιτισμό ε, που έχουμε τώρα, να περάσουμε σε ένα πολιτισμό αγροτών. Τέλος, θα ήθελα να επιθύνω μία έκκληση ε, με την οποία ξέρω πως συμφωνούν πολλοί και να πω ας ξεκινήσουμε εδώ μέσα, στο εστιατόριο εδώ μέσα, στο μπαρ εδώ μέσα, στο πώς τρώμε εδώ μέσα να δείξουμε το καλό παράδειγμα. Ευχαριστώ. Okay, well, we're running a bit... Μάλιστα, ο χρόνος πιέζει. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην ψηφοφορία. Από ό,τι κατάλαβα, έχετε αποσύρει τις προφορικές τροπολογίες και πάμε κατευθείαν συμβαστική τροπολογία 1, γιατί η, η προφορική έχει αποσυρθεί και θα επανεμφανιστεί αργότερα. Οπότε υποβάλλεται η συμβαστική 1 σε ψηφοφορία υπέρ. Κατά. Αποχές Οπότε περνάμε τώρα στην τροπολογία 8. Σχάλτε μόζε. Υπέρ. Κατά. Νομίζω πως θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά άρχη ψηφοφορία ε, επί της τροπολογίας 8. Πέρας. Απορρίπτεται με ισοψηφία 16-16. Τροπολογία 10. Σχαλτεμόζε Άρχεται η ψηφοφορία. Έλα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Δεκτή. 18 με 14. Τροπολογία 11 Σκαλτεμόζε υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβαστική 2. Υπάρχει η προφορική τροπολογία εδώ πέρα που βάζει στην αρχή της συμβαστική 2 το εξή. Τονίζει πως απαιτείται πολιτική βούληση για να εξευρεθούν λύσεις στο ζήτημα αυτό. Ε, υποθέτω πως όλοι συμφωνούν, οπότε τίθεται χωρίς την ε, προσθήκη υπέρ, κατά, δεκτή. Περνάμε τώρα στην 19 Ριούλε υπέρ κατά αποχές 20 υπέρ 20 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ κατά δεκτή. Περνάμε τώρα στην συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Οπότε περνάμε τώρα στην 31. Μπίλεν υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε άρα στην τροπολογία 42 του κ. Σφότ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή, 18 ε, με 14. Τροπολογία 43 της κυρίας Φέντ, Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή και αυτή. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Και τροπολογία 48 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Οπότε ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα για το σχέδιο γνωμοδότησης στο σύνολό του υπέρ. Αρχή ψηφοφορία. The vote's Πέρας. 32 υπέρ. Μία ψήφος κατά. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Οπότε τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες σήμερα. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Εισηγητές και συντάκτες και περνάμε σε μια πρώτη συζήτηση κάποιων γνωμοδοτήσεων που έχουμε. Ε, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση και θα πρέπει να σας παρακαλέσω να είστε σύντομοι γιατί πρέπει να συνεδριάσουν και οι συντονιστές στις 6 ώρα. Οπότε περνάμε απευθείας στην ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση Πιτέλα. Μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως εχμή του δόρατος. Νομίζω είναι για την Επιτροπή Βιομηχανίας. Λοιπόν, ο κύριος Πιτέλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα είμαι λακωνικότατος κύριε Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να ε, διαφωνεί ότι αυτό το σχέδιο δράση μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την χαλεπή στιγμή της ευρωπαϊκής οικονομίας, να συμβάλλει στην ανάκαμψη ε, της ευρωπαϊκής οικονομίας και να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι ένα παράδειγμα πολύ χρήσιμο να έχουμε διαδικτυακές πύλες ε, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προκειμένου να διευκολύσουμε ε, την διασυνοριακή δραστηριότητα και την ίδρυση επιχειρήσεων να ενισχύσουμε την ανάμειξη των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε πληροφορία του κοινού και σκέφτομαι ε, σε ανοιχτέ ε, διακυβερνήσει απέναντι στην βική κράτεια και ε, να βοηθήσουμε όλοι και την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και την ευρωπαϊκή διοίκηση αλλά και τους πολίτες διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε διαδικασίες, στην online πληροφόρηση και επίσης είναι σημαντικό να ζητήσουμε από την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν τη διαλειτουργικότητα στις διάφορες online πλατφόρμες και να χρησιμοποιηθούν υπάρχοντες μηχανισμοί στα κράτη-μέλη ώστε να ενισχύσουμε την ψηφιακή ε, ηλεκτρονική και εσωτερική αγορά. Αυτά και περιμένω τις προτάσεις και παρατηρήσεις από τους κοιόδης συγητές. Ωραία. Μόλις ε, έπιασα τον κύριο Έγκστρομ, ο οποίος από σκιώδης θα γινόταν πραγματικά όρατος, αλλά πριν από αυτό νομίζω πως έχουμε και άλλη μια ομιλήτρια που θα ακούσουμε πριν το τέλος. Λοιπόν, η κυρία Καλνιέτε, ο κύριος Κρόιτσμαν, δεν ξέρω οι υπόλοιποι σκιώδης ηγητές αν θα μιλήσουν. Ο κύριος Έγκστρομ λοιπόν είναι εδώ και μετά θα αντικαταστήσω εγώ τον συνάδελφο που λείπει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε την κυρία Καλνίατε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι και εγώ στο δυνατόν σύντομη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έγγραφο αυτό. Έχω τονίσει πολλές φορές πως πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να μπορέσουμε να, καν, να καταργήσουμε όλα τα εμπόδια στην ενιαία αγορά. Οι έρευνες δείχνουν πως ακόμα δεν ε, χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δεν υπάρχουν ακόμα ε, σελίδες όπου μπορούν να ευρεθούν οι ε, υπηρεσίες. Να αναφέρω το Solvit Europe. Δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες, γι' αυτό φταίμε εμείς, αλλά και τα κράτη-μέλη φταίνε εν μέρη. Θα ήθελα λοιπόν να στηρίξω την έκκληση του να υπάρξει ένα πόρταλ για επιχειρήσεις και να υπάρχει μία, ένας ενιαίος κατάλογος σημείων επαφής για να διευκολυνθεί η δουλειά των επιχειρήσεων και η συνεργασία επίσης. Ελπίζω να το επιτύχουμε αυτό στο μόνο για το εμπόριο έχουμε μεγάλο δυνα... υπάρχουν πολλές δυνατότητες εδώ πέρα και ελπίζω πως ε, οτιδήποτε μυρίζει προστατευτισμό δεν θα πρέπει να επιτραπεί. Θα καταθέσω πολλές προτάσεις και είμαι σίγουρη πως η Επιτροπή μας θα εγκρίνει ένα ε, καλό και ισορροπημένο σχέδιο και θα προωθεί έτσι ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριος Κρόιτσμαν. Νομίζω δεν είναι εδώ. Λοιπόν, ο κύριος Έγκστρομ. Ευχαριστώ. Νομίζω πως ε, το σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Πιτέλα είναι πολύ λογικό. Συμφωνώ. Και δεν έχω κάποια ιδιαίτερη παρατήρηση. Ναι, ναι, μια χαρά μου φαίνεται. Ε, Ευχαριστώ. Ο κύριος Κότσουσνικ επίσης μου ζήτησε να συγχαρώ και εγώ τον εισηγητή. Του αρέσει ιδιαίτερα η παράγραφος 2 εκεί όπου μιλάτε για την διευκόλυνση κινητικότητας και τη μείωση της γραφειοκρατίας, κάτι το οποίο τον αφορά ιδιαίτερα. Και βεβαίως καλωσορίζουμε το ότι τονίζεται τη σημασία των ηλεκτρονικών προμηθειών. Αυτό το ανέφερε και η έκθεση Ριούλε. Και νομίζω πρέπει να τον ισχύσουμε και ειδικά το σημείο που αναφέρει τα πιθανά ωφέλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την πρόσβαση στις ε, κρατικές υπηρεσίες. Οπότε κάποιες τροπολογίες θα υπάρξουν εκεί πέρα για να προσθέσουμε νομίζω στην πολύ καλή σας έκθεση. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Θέλει κάποιο άλλο να μιλήσει. Ο κύριος Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν ο Αντιπρόεδρος της Βουλής ε, ανέθεσε στον κύριο Πιτέλα τη γνωμοδότηση, σκέφτηκα πως θα έχουμε μια έντονη ανταλλαγή απόψεων. Βεβαίως είναι καλή ε, η γνωμοδότηση, αλλά νομίζω πως θα έπρεπε να τονίσουμε το ότι μειώνουν οι πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τα γραφειοκρατικά εμπόδια και το κόστος και θα πρέπει άρα να υπάρξει μια βελτίωση προς αυτή την έκθεση. Αναφέρεται στην έκθεση, πρέπει να τονιστεί νομίζω δεύτερον. Υπάρχουν αυτά τα Solvit και το Europe, τα Portal, τα πανευρωπαϊκά και θα μπορούσαμε να τα τονίσουμε. Τρίτον, Μπορούμε βέβαια να σκεφτούμε το τι μπορεί να γίνει με περαιτέρω σύνδεση των διαφόρων δικτύων. Ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν ευκολότερη και απλούστερη πρόσβαση σε πληροφορίες, σε εργαλεία, δυνατότητες με ένα κεντρικό αποτελεσματικό δίκτυο και έτσι θα ενισχυθεί η κινητικότητα και η δυσναριακή δραστηριότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ιδιαίτερα. Επίσης βρίσκω θετικό το ότι ο κύριος Πιτέλα έχει αναφέρει το, τη μία ε, υπηρεσία στην οποία μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτες, αλλά βεβαίως θα πρέπει να τονίσουμε πώς θα πρέπει να βελτιωθούν αυτές οι υπηρεσίες και να εφαρμοστούν σωστά από τα κράτη-μέλη. Εδώ πέρα είχαμε και την υπηρεσία, νομίζω, για την οδηγία, για τη, τη συζήτηση για την οδηγία περί και υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες που θα πρέπει να από όσα Έχω και άλλα να πω κύριε Πρόεδρε, αλλά νομίζω πως αυτά αρκούν για την ώρα και βεβαίως ε, αναμένω τη συνεργασία την περαιτέρω με τον κύριο Πιτέλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, ξέχασα και εγώ να σας ε, ε, απευθύνω το λόγο με αυτόν τον τίτλο. Συγγνώμη. Κύριε Βίλντε, θέλετε και εσείς να προσθέσετε κάτι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βίλτε, Wilde, το ίδιο είναι για μένα. Είμαι ελαστική στην προφορά του όνοματό μου. Συμμεριζόμαστε πλήρω τις προτεραιότητε του συντάκτη τη γνωμοδότηση, γιατί ανταποκρίνονται στις δράσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ιδιαίτερα σε ό,τι φορά τον περιορισμό τη γραφειοκρατίας και την, ε, το διασυνοριακό χαρακτήρα των υπηρεσιών κυρίως με τη χρήση επιγραμμικών υπηρεσιών. Όσο περισσότερες επιγραμμικές και ψηφιακές διαδικασίες έχουμε, τόσο πιο πολύ περιορίζουμε την γραφειοκρατία. Επίσης, στενιζόμαστε τη σημασία που έχει η διαλειτουργικότητα στις ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες. Έχουμε το PEPOL, ένα σχέδιο που αναφέρεται, αν δεν κάνω λάθος, στη γνωμοδότηση, την πρωτοβουλία PEPOL και η και αυτές θα βελτιώσουν τις δημόσιες προμήθειες ε, online. Δεν αναφέρθηκε φέρθηκε τους υπόψη το θέμα της συμμετοχής γιατί το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας στην λήψη αποφάσεων διακυβέρνησης και να εμπλέξει περισσότερο του πολίτες και τις επιχειρήσεις στη διαδικασία λήψη αποφάσεων κάποιες μορφές για το ότι δεν περιλαμβάνονται τα ηλεκτρονικά προσόντα, ηλεκτρονικές δεξιότητες. Είναι πολύ σημαντικές και τις καλύπτουμε σε άλλο σημείο, αλλά ε, με ευρύτερη έννοια τις καλύπτουμε και εδώ αυτές οι ηλεκτρονικές δεξιότητες. Άλλωστε περιλαμβάνονται και στο ψηφιακό πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Ξαναδίδω το λόγο στον Αντιπρόεδρο Πιτέλα για μια ανακεφαλαίωση και για να μας επιβεβαιώσει και το χρονοδιάγραμμα. Αρκεί και μισό λεπτό να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, τον Πρόεδρο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρετε ότι δεν είμαι τυπολάτρης, είμαι άνθρωπος της ουσίας παρά του τύπου, γι' αυτό και δεν με ενδιαφέρουν και οι τίτλοι. Ο κύριος Σβάπ ήταν πολύ ε, ευγενικός και στοργικό, ε, υπεθυμίζοντας τον τίτλο μου. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ως προς τους στόχους που θεσπίσαμε. Έχουμε ένα σχέδιο γνωμοδότης, αν υποβληθούν τροπολογίες θα τις λάβω υπόψη. Κοινό μας στόχος πάντως είναι να γίνει η Ευρώπη όσο πιο διαφανής γίνεται και όσο πιο κοντά ε, προς τον Ευρωπαίο πολίτη γίνεται. Να εξασφαλίσουμε πρόσβαση του πολίτη σε όσο περισσότερα δεδομένα γίνεται, να αυξήσουμε την απασχόληση, να ανακάμψει η οικονομία μας και να δημιουργήσουμε μια γνήσια δημοκρατία. Γιατί πολλές φορές μας προσάπτουν ότι είμαστε οι προασπιστές της γραφειοκρατίας. Αυτό τον ε, δυσμενή τίτλο θα πρέπει πραγματικά να τον διαψεύσουμε, προβάλλοντας τη δημοκρατία και την καταπάρα περιορίζονται στην γραφειοκρατία. Σα ευχαριστώ. Και το χρονοδιάγραμμα 27 Οκτωβρίου λίγη η διορία για τις προθεσμίες, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Εξέταση τροπολογιών και ψηφοφορία 26 Νοεμβρίου, ώστε να πάει στην Ήτρε που θα ψηφίσει στις 19 Δεκεμβρίου και στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο του 2012. Και μάλλον θα είστε εκεί για να λάβετε το λόγο κύριε Σιγητά. Σας ευχαριστώ. Τώρα ψάχνουμε ακόμη το χαμένο μας εισηγητή, γιατί μας διέφυγε ο κύριος Φόξ, ο συντάκτης γνωμοδότη. Φαντάζομαι θα επανέλθει σύντομα να κάνω μια απογραφή των σκιωδών εισηγητών αυτή τη σημαντική αιτήσια γνωμοδότηση για την, της μάλλον για την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος, Σβάπ από το ΕΛΚ, η κυρία Γκέπχαρντ από τους Σοσιαλιστές, ο κύριος Μπουζόη, κάποιος άλλος από την Άλντε, ουδής, η κυρία Ρούλε, ο κύριος Άγκστ Κύριε κυρία Ρούλε. Άλλος κανείς, άλλοι εθελοντές για την γνωμοδότηση του κύριου Φόξ. Έχουμε και τον Τέρ Μπρόνς. Με ενημερώνουν ότι θα καταφτάσει ένα πάει στιγμή ο κύριος Φόξ. Just while we're doing that, then, just me talk to you about the timetable. Στο όσο αναμένουμε τον εισηγητή μας, ε, να σας υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμά μας. Το χρονοδιάγραμμα λοιπόν. Πολύ πιστικό, γιατί η αρμόδια επιτροπή ΕΚΟΝ θα ψηφίσει στις 22 Νοεμβρίου Οπότε οι δικές μας τροπολογίες θα πρέπει να εξεταστούν και να ψηφιστούν στις 21 Νοεμβρίου. Φαντάζομαι ο κύριος Φόξ θα προτείνει με έξυπνο τρόπο, θα προβάλλει τις ε, τροπολογίες μας στην εικόνα ώστε να ληφθούν υπόψη. Άλλες διορίες. Η διορία για την υποβολή τροπολογιών λήγει στις 26 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι. Ο κύριος Φάμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για τον κανονισμό. Να πω πως οπωσδήποτε δεν είχαμε επιθυμία να καταθέσουμε τροπολογίες στις συμβιβαστικές τροπολογίες. Και ούτε θέλαμε να ενοχλήσουμε τους σοσιαλδημοκράτες ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Απλά θα ήθελα να γνωρίζω εάν οι πρόεδροι, χωρίς να το γνωρίζω εγώ, κατέληξαν σε έναν άλλο κανονισμό. Εάν δεν έχει γίνει αυτό, όλα είναι εντάξει. Αυτό το οποίο ήθελα είναι απλά να έχουμε την δυνατότητα με τις τροπολογίες, τις συμβαστικές, να επιτρέψουμε χωριστές ψηφοφορίες σε κάποια προχωρημένη φάση. Νομίζω πως μπορούμε να τα καταφέρουμε, νομίζω πως το θένε και οι συντονιστές. Πρόκειται απλά για ερμηνεία του κανονισμού των Επιτροπών. Εγώ είπα ότι θα ακολουθήσω τις πολιτικές ομάδες και τους συντονιστές. Ό,τι συμφωνήσουν θα το σπαστώ. Ε, δεν παραπονέθηκα εγώ για τις ψηφοφορίες κατά τη Να, να πω και εγώ λίγο κάτι. Κοιτάξτε, οι περισσότερες χωριστές ψηφοφορίες είναι έτοιμα του ΕΛΚ, οπότε νομίζω πως δεν έχουμε κι εμείς ε, κανένα ενδιαφέρον να αλλάξει η διαδικασία, άρα δεν υπάρχει και λόγο νομίζω να μιλάμε. Ελπίζω έτσι. I mean, I don't think as far as... Ε, από ό,τι μου φαίνεται η γραμματεία σχετικά με τη διαδικασία δεν μας εμποδίζει τίποτα από το να ζητάμε ε, στην Επιτροπή ξεχωριστές ψηφοφορίες για συμβιβαστικές τροπολογίες, αλλά όχι για συμβιβαστικές στην Ολομέλεια. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία γιατί μερικές φορές στην Ολομέλεια αντιπροσωπεύουν σημαντικές συμφωνίες ανάμεσα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο, οπότε προφανώς δεν μπορούμε εμείς να αλλοιώσουμε το τελικό αποτέλεσμα πριν την ψηφοφορία αλλά για τις επιτροπές θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι εφόσον συμφωνούν και οι υπόλοιπε πολιτικές ομάδες και νομίζω ότι η άποψη της κυρίας Γκέπχαρτ είναι σωστή. Σε σκληρές διαπραγματεύσεις είναι αλήθεια ότι την τελευταία στιγμή καταλήγουμε σε συμβιβασμούς, αλλά οι επιτροπές αν θέλουν να κάνουν αλλαγές το κάνουν, δικαίωμά τους επαφίεται στη λογική, αν θέλετε, των ομάδων που καταθέτουν τις προτάσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα δεδικασμένο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αν και ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να πιστεύει κάτι το διαφορετικό. Κύριε Φόξ, καλώς ήρθατε. Ο άλλος Φόξ έχει πρωτοσέλιδα στην πατρίδα σας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, παρότι το κόμμα μας δεν είναι ενθουσιασμένο, θα μας μιλήσετε για τον πολιτική ανταγωνισμό. Ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ στην κατάλληλη στιγμή. Έπρεπε αμέσως μετά τις ψηφοφορίες να πάω κάπου αλλού. Λοιπόν, για την πολιτική ανταγωνισμού, την έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού. Είναι, θα έλεγα, προϊόν και ανάπτυγμα της ε, εσωτερικής αγοράς, όχι μόνο για τον σωστό ανταγωνισμό, αλλά και για τις επιλογές προς τον καταναλωτή. Πρέπει να συγχωρούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δουλειά της εδώ σχετικά με, την, με το θέμα της επιβολής των κανόνων. Είναι η 40η επέτειος της έκθεσης και θα ήθελα η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς να συγκεντρώσει την προσοχή της στη διαφάνεια και στις επιλογές προς τους καταναλωτές. Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να εμείνουμε σε πέντε συγκεκριμένους τομείς. Διαφάνεια στις τιμές, ε, προσπάθεια να διασφαλίσουμε την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, την, ε, τον έλεγχο των τιμών της ενέργειας και τις αρνητικές συνέπειες ε, της, ε, του μη σεβασμού των κανόνων του ανταγωνισμού. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά, αλλά κάποια από αυτά μπορούμε. Η αυξημένη διαφάνεια δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να αξιολογεί στην αγορά και να αναλύσει τις δομές των τιμών αυξάνει τον ανταγωνισμό, ανοίγει τις αγορές, αυξάνει τις επιλογές για τους καταναλωτές, ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους. Παράδειγμα, όταν αυξάνεται το κόστος το χονδρικό της ενέργειας, αυξάνεται υπερβολικά και η λιανική τιμή αλλά όταν πέφτει η χονδρική τιμή ελάχιστα μειώνεται η λιανική. Αυτό είναι απαραδεκτό και νομίζω ότι η αυξημένη διαφάνεια στις αγορές θα βοηθήσει να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο και σε ποιο βαθμό είναι δικαιολογημένο. Μπορούμε να ενθαρρύνουμε λοιπόν πολλά από αυτά τα θέματα αν κάνουμε συγκεκριμένες πρακτικές προτάσεις τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν για να δώσουν την δυνατότητα στους καταναλωτές να λειτουργήσουν σωστά. Θα συνεργαστώ λοιπόν και με τους Κιώδης και να προωθήσουμε τις συγκεκριμένα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε και κύριε Κύριε Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Φόξ πράγματι ανέφερε τα σημεία τα οποία θεωρεί σημαντικά. Μπορώ να συμφωνήσω μαζί του σε μεγάλο βαθμό, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για το ότι ε, μπορέσαμε να προσαρμόσουμε το πρόγραμμά μας με αυτό της ε, κατά κύριο λόγο αρμόδιας Επιτροπής Οικονομικών και εξάλλου δεν έχει νόημα για μια έκθεση του 2009 να εκφέρουμε γνώμη το 2011. Θα πρέπει να γίνονται τα πράγματα εγκαίρως. Και νομίζω το ότι ψηφίζουμε μία μέρα πριν την Επιτροπή Οικονομικών μας δίνει τη δυνατότητα να αναφέρουμε αρκετά πράγματα. Γι' αυτό το οποίο είπε ο κύριος Φόξ θα ήθελα εγώ να πω μόνο ένα ζήτημα, αυτό το οποίο αναφέρεται στο σημείο 6 του καταλογού του και εγώ χαιρετίζω την απόφαση των Υπουργών για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, αλλά δεν είναι το μόνο μέτρο ανταγωνιστικότητας. Είναι θετικό, αλλά όχι το η μόνη θετική απόφαση. Για ε, μπορώ ε, έτσι να το στηρίξω. Επίσης, για το θέμα της διαφάνειας του κυρίου Φόξ, να αναφέρω πως ο καταναλωτής συχνά αποφάσεις ε, περί δικαίου του ανταγωνισμού της ε, Κομισιόν δεν μπορεί να τις παρακολουθήσει και το τονίζει αυτό και η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων και είναι βεβαίως ζήτημα αποτελεσματικότητας και διαφάνειας των προστήμων. Οπότε θα πρέπει και οι αρχές επιβολής των προστήμων να περιλαμβάνονται στην απόφαση και να επανεξετάζονται από καιρού καιρών. Και εδώ πέρα παίζει ένα ρόλο το κατά πόσον μπορούν να πάνε τα χρήματα αυτά του προστίμου και στους καταναλωτές οι οποίοι έχουν πληγεί από ένα καρτέλ. Και είναι σημαντικό επίσης το ότι μπορούμε να παρέμβουμε εγκαίρως στο έργο της Επιτροπής Οικονομικών. Σας ευχαριστώ κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ. Ίσως η Επιτροπή Οικονομικών θα μπορούσε να στέλνει αυτά τα πράγματα νωρίτερα για να μην υπάρχει αυτή η χρονική πίεση. Γιατί βεβαίως ε, και εμείς θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά εδώ πέρα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φόξ για το σχέδιο γνωμοδότησής του, το οποίο βρίσκω πάρα πολύ θετικό. Και ακριβώς αυτά τα θέματα, διαφάνεια των τιμών δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και μπορούμε να φέρουμε και άλλα παραδείγματα στα οποία θα θέλαμε να καταθέσουμε τροπολογίες όπως η περιαγωγή, αλλά και άλλα. Επίσης, θετικό βρίσκω το σημείο 3 που έχετε, όπου μιλάμε για την διαφάνεια, για την διατροφική αλυσίδα για να γνωρίζουμε πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Γιατί ακούμε πάντα τον καυγά μεταξύ γεωργών που λένε πως εμείς παίρνουμε ψίχουλα για τα προϊόντα μας και του καταναλωτή ο οποίος πληρώνει πάρα πολύ για τα τρόφιμα. Εάν δει κανείς πράγματι τη διαφορά στη μέσα, ρωτιέται πού πάνε τότε τα λεφτά. Και το να έχουμε αυτή την πληροφόρηση θα ήταν καλό. Και να αναφέρω άλλη μια πτυχή, την ποιότητα των προϊόν, προϊόντων που δεν αναφέρατε, αλλά επίσης παίζει σημαντικό ρόλο. Αλλιώς, πράγματι είμαι σίγουρη πως θα έχουμε καλή συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ. Χριστιαν Μπουζόη, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Φόξ για το σχέδιο γνωμοδοτησή του που είναι πάρα πολύ σημαντικό και τονίζει κάποια στοιχεία για την ανάπτυξη μιας ιστορικής αγοράς με ανταγωνισμό. Καλωσορίζω την αναφορά στον τομέα της ενέργειας όπου θα πρέπει να διασφαλιστεί ο ανταγωνισμός για να υπάρχει μια πραγματική ιστορική αγορά ενέργειας. Χάρηκα ιδιαίτερα για το ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν καταργήσει τις ε, τιμές ε, οι οποίες ήταν ρυθμισμένες και αυτό είναι σημαντικό για να υπάρξει ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Επίσης, ορίζει να αφορά στο σύστημα ευρεσιτεχνίας της Ένωσης που θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον τομέα τον φαρμακευτικό, παραδείγματος χάρη, αλλά και για άλλους. Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω κάτι για το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων που δεν αναφέρεται στο σχέδιο γνωμοδότησης θεωρώ αυτό το προσωρινό πλαίσιο και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διατηρηθεί ενισχύ μέχρι το τέλος του έτους πάρα πολύ ρεαλιστική. Αυτό ήταν απαραίτητο για να διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να συνεχίσουν οι τράπεζες να εκπληρώνουν το ρόλο τους, δηλαδή την πίστοση στην πραγματική οικονομία. Και πράγματι η ανάκαμψη πέρσι ήταν πάρα πολύ αργή και βεβαίως ε, τώρα είμαστε ακόμη πάρα πολύ κοντά σε κίνδυνο ύφεση. Πρέπει να το έχει αυτό υπόψη η Κομισιόν, να έχει μια ρεαλιστική προσέγγιση, αλλά να εξετάζουμε και άλλε λύσει, γιατί δεν μπορούμε βεβαίω να διατηρούμε αυτό το ενδιάμεσο πλαίσιο σε ισχύ. Τέλο, χαιρετίζω τη συμφωνία μεταξύ Βίζα και Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πολυμερή τέλη χρέωση και το επίπεδο μειώθηκε σε 0,2%. Νομίζω λοιπόν πως είναι θετική αυτή η εξέλιξη, καθώς έτσι θα είναι ευκολότερο για τους καταναλωτές να πληρώνουν με κάρτα όταν ψωνίζουν χωρίς ε, επιπρόσθετο κόστος. Ε, θεωρώ πως πραγματικά μπαίνουμε σε ε, μια κατάσταση φυσιολογική, γιατί μιλάμε για ψηφιακή ατζέντα, ηλεκτρονικό εμπόριο και από την άλλη αντιμετωπίζουμε περιορισμούς στις ηλεκτρονικές συναλλαγές λόγω του τέλους αυτού που επομίζεται ο καταναλωτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρούλε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το ότι επικεντρώθηκε σε λίγα πράγματα γιατί νομίζω πως έτσι είμαστε πιο αποτελεσματικοί ως Επιτροπή εάν δεν ασχολούμαστε με τα πάντα. Επίσης αυτό το οποίο ανέφερε η κυρία Γκέμπχαρτ, το roaming και αυτό πρέπει να τα αναφέρουμε εδώ πέρα γιατί νομίζω είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών. Αλλιώς αυτά τα οποία έχετε εσείς εδώ πέρα ε, ενέργεια και αλυσίδα τροφίμων. Σημαντικά εκεί πέρα δεν υπάρχει διαφάνεια. Επίσης τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις μπορούμε να το συμπληρώσουμε, αλλά νομίζω πως έχουμε βρει τα σωστά σημεία και πράγματι σας στηρίζω. Καλά σας ευχαριστώ. Ως πρόεδρος θα ήθελα να πω ότι ο συνδυασμός με την πρόταση για την διαφάνεια των τιμών είναι πολύ σημαντικός να δούμε και τις επιδόσεις σε ό,τι αφορά τις, κα, τους καταναλωτές και τις τιμές, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις τιμές ε, βασικών αγαθών μεταξύ των χωρών, κάτι που δείχνει πραγματικά έλλειψη μιας αποτελεσματικής αγοράς για τους καταναλωτές. Αυτό ίσως θα ήθελα να το λάβει υπόψη η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και να κοιτάξει αυτούς τους δείκτες τιμών γιατί ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός είναι σημαντικός και για τον καταναλωτή. Θα το συζητήσουμε και με τους συντονιστές, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να καλέσουμε μια μέρα την Επιτροπή να έρθει να μας μιλήσει. Γιατί ο Επίτροπος Ανταγωνισμού θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο και για τους καταναλωτές. Ίσως θα πρέπει να το αφήσουμε για το επόμενο χρόνο όμως αυτή τη συνάντηση. Ε, δεν ξέρω, ελάχιστο χρόνο μα έχει μείνει. Κυρία Μπρόγκ, θέλετε να το σχολιάσετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την πρόταση. Είναι ευαίσθητη στα θέματα της εσωτερικής αγοράς και της ενέργειας και της διαφάνειας της τροφιμικής αλυσίδας θεωρούμε πολύ σημαντική την σημασία την οποία δίνει στην ε, προσπάθεια για επίτευξη διαφάνειας. Δεν έχουμε περαιτέρω σχόλια να κάνουμε σε αυτή τη φάση και περιμένουμε τις τροπολογίες. Uh, um, Κύριε Φόξ, λοιπόν μας έχετε δώσει το χρονοδιάγραμμα, μπορείτε να κλείσετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους και όλες για τη συνεισφορά τους. Παρατήρησα τα σχόλιά σας για τα πίνακες αποτελεσμάτων της αγοράς και των καταναλωτών. Άκουσα αυτά τα οποία είπε και η κυρία Ρούλε για, την, για το roaming στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Αλλά πέραν αυτό νομίζω ότι η συζήτηση ήταν αρκετά επικοδομητική. Λοιπόν, εντάξει, τώρα κανονικά θα συζητούσαμε το επόμενο θέμα, το οποίο αφορά την έκθεση Μακλάρκιν για την πρόοδο της διαδικασίας της Μπολόνια. Έρχεται η κυρία Μακλάρκιν. Ήρθε τη σωστή στιγμή λοιπόν. Έχουμε και τον κύριο Τάισεν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για μια έκθεση που ανήκει στην Επιτροπή ε, Πολιτισμού και Εκπαίδευσης για τα ευρωπαϊκά όργανα και την πρόοδο στη διαδικασία της Μπολόνια έχει κάτι το οποίο συνδέεται θα έλεγα με την γνωμοδότηση που μόλις ψηφίσαμε κιόλας και γι' αυτό και Μακλάκιν σου δίνω το λόγο για να παρουσιάσει τη γνωμοδότησή σου. Ξέρω ότι ήταν δύσκολη ημέρα αλλά σε καλωσορίζουμε για μια ακόμη φορά. Πρόεδρε, ο χρονισμός ήταν ο κατάλληλος. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Όπως ξέρετε, η διαδικασία της Μπολόνια είναι ένα τμήμα μιας μακροπρόθεσμης και φιλόδοξης διαδικασίας για ένα ευρωπαϊκό χώρο παιδείας που αφορά και τα πανεπιστήμια και τους επαγγελματίες. Συμμετέχουν τα πιο δυναμικά πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ευρώπη αν θέλουμε πράγματι να ανταγωνιστούμε την Κίνα και την Ινδία που έχουν φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Πρέπει οι νέοι να μπορέσουν να αναπτύξουν και την απασχολησιμότητά τους και νομίζω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα συγκρίσιμο και συμβατό σύστημα που να βελτιώνει την κατάσταση. Υπογραμμίζουμε την έρευνα, την καινοτομία, κάνουμε τα πανεπιστήμια μας πιο ανταγωνιστικά και υπογραμμίζουμε την, τον στενό δεσμό της διαδικασίας της Μπολόνια και της επαγγελματική κατάρτισης. Για όλα αυτά λοιπόν ζητάμε από την Επιτροπή να βελτιώσει τη δυνατότητα μεταφοράς διδακτικών μονάδων και να χρησιμοποιηθεί σαν μέσο αναγνώρισης ακριβώς των ικανοτήτων των επαγγελματικών. Σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι η επόμενη 5η 12η Μεσημβρινή και θα ψηφίσουμε στις 22 Νοεμβρίου θα έλθω σε επαφή με τους σκιώδεις για να έχουμε μια συνάντηση πριν από αυτή την ψηφοφορία και να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην μεθεπόμενη ολομέλεια του Στρασβούργου. Περιμένω με αγωνία τα σχόλιά σας. Έχουμε μαζί μας την κυρία Λεγκρίπ, κυρία Βερνιολίπη και την κυρία Γκέπχαρτ. Και η κυρία Ρούλε επίσης, αν θέλει μπορεί να πάρει το λόγο. Ωραία, πρώτα κυρία Λεγκρίπ. Ευχαριστώ. Μιλούμε και πάλι για την κινητικότητα. Πώς αντιευκολύνουμε διευκολύνουμε την κινητικότητα των συμπολιτών μας. Ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο και της εσωτερικής αγοράς, αλλά και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Είμαστε φυσικά, όπως είδατε, υπέρ ε, της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και είδατε με τι μεγάλη πλειοψηφία εγκρίναμε την προηγούμενη έκθεση της κυρίας Είμαι κινηματογραφόφιλος, γι' αυτό επ' ευκαιρία της ε, γνωμοδότησης ε, θυμήθηκα δύο σημαντικές ταινίες γαλλικές, το Λομπέρζο Σπανιόλ, το ε, Οσπιανικό Παδοχείο και την ε, Ρωσική Κουκλέλα που Περούς είναι δύο ταινίες που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό και που κυκλοφόρησαν ευρέως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματικά αυτές οι δύο γαλλικές ταινίες ε, δείχνουν και με εικόνα και με ήχο και με ε, τους ηθοποιούς αυτούς την ανάγκη αύξησης και βελτίωσης της κινητικότητας ε, των φοιτητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ με την ε, συντάκτρια της γνωμοδότησης και με την έμφαση που δίνει στα διάφορα σημεία. Δεν πρόκειται να απαριθμίσω όλα τα σημεία της συμφωνίας μας. Είναι πολλά και σημαντικά. Πάντως είμαι στη διάθεση της ε, εισηγητριάς μας, της συντάκτηρας γνωμοδότησης, για να επικεντρωθούμε σε δύο-τρία σημεία συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, θα ήθελα στη γνωμοδότηση αυτή να κάνουμε μια του προγράμματος έρασμος. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με το θέμα αυτό, αλλά δεδομένη της επιτυχίας του προγράμματος αυτού και του μεγάλου αριθμού των φοιτητών, το 2010 για παράδειγμα είχαμε 2.200.000 ε, φοιτητές που έλαβαν υποτροφίες από το Έρασμος. Τεράστια επιτυχία, γιατί λοιπόν να μην αποτίσουμε φοροτιμή στο πρόγραμμα αυτό και δεδομένη τη σπουδαιότητα που είχε το πρόγραμμα έρασμο, καλό θα ήταν να συνεχίσει να χρηματοδοτείται με σημαντικά κονδύλια. Να εξασφαλίσουμε βιωσιμότητα αυτών των κονδυλίων, και, γιατί όχι και αύξησή τους, αν και αυτό θα ήταν υπερβολικά φιλόδοξο. Πάντως, ε, ε, επί τη ευκαιρία της γνωμοδότης, καλό θα ήταν να διατρανώσουμε την υποστήριξή μας στο πρόγραμμα Έρασμος. Ίσως ε, με την ευκαιρία της γνωμοδότησης θα μπορούσαμε να προτείνουμε και την λήψη υπόψη στο σύστημα Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Δακτικών Μονάδων, τη λήψη υπόψη και των πρακτικών ασκήσεων που γίνονται στα πλαίσια των σπουδών, στο εξωτερικό. Να ληφθούν υπόψη και αυτά τα στάσεις και αυτές οι πρακτικές ασκήσεις, γιατί και οι, οι πρακτικές ασκήσεις αποτελούν τμήμα του προγράμματος σπουδών, γιατί να μην συμπεριληφθούν και αυτές λοιπόν στο σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων. Και κάτι άλλο, να ενισχύσουμε την κατάρτιση σε όλα τα στάδια των σπουδών, και στην αρχή και στη μέση και προς το τέλος των σπουδών. Έτσι θα βελτιωθεί η κινητικότητα, γιατί σε ορισμένες χώρες ε, υπάρχει υποαπορρόφηση των υποτροφιών του προγράμματος Έρασμος. Γιατί λοιπόν να μην ενημερώσουμε καλύτερα τα πανεπιστήμια, τα κράτη-μέλη και όλες τις οργανώσεις για τις δυνατότητες που υπάρχουν, ώστε να εκταμιεύονται όλες οι υποτροφίες του προγράμματος Έρασμος. Αυτά, εν ολίγης, τα σημεία που θα ήθελα να επισημάνω και θα υποβάλω και κάποιες τροπολογίες. Πάντως, ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μακλάρκιν και τη συγχαίρω θερμά για την πολύ αξιόλογη της γνωμοδότηση. Uh, Ευχαριστούμε κύριε Λεγκρίπ. κύριε Γκέπχαρτ. Και κυρία Βερνιό θα, σίγουρα θα ενδιαφερθεί για το θέμα αυτό και θα υποβάλει σχόλιο. Κύριος Μπουσόη. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και χαίρομαι για το ότι έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε ξανά με την κυρία Μακλάρκιν όχι μόνο στην αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, αλλά και στη διαδικασία της Μπολόνιας και θεωρώ πως υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο εκθέσεων. Ακόμα και αν το σύστημα δεν λειτουργεί πάντα τέλεια, λόγω της άνησης εφαρμογής, πρέπει να παραδεχτούμε πως η διαδικασία της Μπολόνιας ενίσχυσε την κινητικότητα των φοιτητών Επίσης πρέπει να έχουμε ευρύτερη αντικειμενική εικόνα για την εφαρμογή της διαδικασίας Μπολόνιας, να ξέρουμε που δεν έχει εφαρμοστεί επαρκώς για να αναλάβουμε δράση. Ένα άλλο σημείο το οποίο θα υποστήριζε ευχάριστος είναι η κινητικότητα των ερευνητών, το έχουμε ήδη τονίσει και στην έκθεση της Λάρα ακόμη για την έρευνα και την καινοτομία και νομίζω πως μπορεί να το επιτύχει αυτό η διαδικασία της Μπολόνιας. Για να επανέλθουμε στη σχέση μεταξύ αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και διαδικασίας Μπολόνιας, νομίζω πως θα πρέπει να ενισχυθεί η σχέση. Καλό είναι οι φοιτητέ να σπουδάζουν στο εξωτερικό, αλλά βλέπουμε να υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση για την αναγνώριση των προσόντων που θα αποκτήσουν εκεί. Πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων οι φοιτητέ για το τι ευκαιρίε θα έχουν και για το εάν τα προσόντα του θα αναγνωρίζονται όταν επιστρέψουν στη χώρα του ή σε άλλο κράτο μέλο. Έχω ακούσει περιπτώσεις που είναι δύσκολο να αναγνωρίσουν τα μαθήματα που έδωσαν οι φοιτητέ και έπρεπε να τα περάσουν δύο φορές. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία όσον αφορά το περιεχόμενο ε, των σπουδών για να γίνουν ευκολότερες οι μεταφορές διδακτικών μονάδων. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την κυρία Μακλάρκιν. Ευχαριστώ κυρία Ρούλε. Έχετε τον λόγο. Καλώς όριζω και την κυρία Βανιό, η οποία νομίζω μπορεί να ολοκληρώσει. Μιλήστε εσείς όμως πρώτα. Ευχαριστώ αντικαθιστώ και την Έμιλη Τούρνεν η οποία απουσιάζει σήμερα και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια θεωρώ πώς θα πρέπει πράγματι να δοθεί βάρος στην ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη μια ενός ευρέως φάσματος δεξιοτήτων ε, ε, και είναι σημαντικό αυτό για τον στόχο της αηφόρου ανάπτυξης, άρα θα πρέπει επίσης να δούμε ποια είναι και η εμπειρία που έχουμε στα κράτη-μέλη με τη διαδικασία της Μπολόνιας. Αυτή διαφέρει γιατί είναι διαφορετική και η εφαρμογή. Οπότε θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που θα βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή των κρατών μελών και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μπουσόη και η κυρία Λεκρύπ για το πρόβλημα της μεταφοράς και της αναγνώρισης των μαθημάτων και στο δικό μου το κράτος και ασκείται κριτική σε αυτό ότι οι φοιτητέ ευχαρίστως θέλουν να πάνε στο Εράσμους αλλά μετά δεν ξέρουν τι θα γίνει με τα μαθήματά τους εκεί πέρα αν θα αναγνωριστούν και αν θα τους χρησιμεύσει. Και οι ταινίε που αναφέρατε ε, είναι πάρα πολύ ωραίες. Πράγματι τις έχω δει και στα γερμανικά και Πρόκειται νομίζω για μια ποιοτική ανάλυση που θα πρέπει να κάνουμε σε διαδικασία της Μπολόνιας μέσω των κρατών Μπολόνια, να έχουμε πληροφορίες που λειτουργεί σωστά και που υπάρχουν προβλήματα. Thank you very much. Mrs. Συγγνώμη που απουσίασα, λέει κυρία Βερνιό. δεν υπολόγισα καλά το χρόνο. Ελπίζω ότι καθυστέρηση, θα εκμεταλλευόμουν την καθυστέρηση. Εν πάση περιπτώσει, συγχαρητήρια κυρία Μακλάρκιν. Γενικώ είναι καλή η γνωμοδότησή σα. Έχουμε και ε, ούτω ή άλλω περιορισμένη έκταση για τι γνωμοδοτήσει. Πάντω τα καταφέρατε και επισημάνατε πολλά θέματα. Τώρα για τι παραγράφου 1 και 3. Τα προγράμματα που επισημαίνετε και το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί θα πρέπει να διευκρινίσουμε το, το σύνδεσμο της, ε, της διαδικασίας Μπολόνιας που περιλαμβάνει 49 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το θέμα του, του προγράμματος ποδρών, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Δακτικών Μονάδων και την πιστοποίηση των πτυχίων. Νομίζω ότι γενικά το σύστημα λειτουργεί καλά, αλλά δεν είναι μόνο θέμα εναρμόνισης ε, των καταρτήσεων και των επαγγελματικών προσόντων, είναι θέμα εξυγχρονισμού της νοοτροπίας θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε το ρόλο των θεσμικών οργάνων. Ε, δεν θα πρέπει βέβαια να είμαστε υπερβολικά απαιτητικοί απέναντι στα πανεπιστήμια γιατί ίσω προκαλέσουμε τη δυσαρέσκεια του. ή να είμαστε υπερβολικά επιτακτικοί, αλλά καλό θα ήταν ε, να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια για να διευκολύνουμε την αναγνώριση και την κινητικότητα μεταξύ των φοιτητών. Γιατί τα προγράμματα σπουδών είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ μια χώρα και άλλη, ακόμη και μεταξύ μια σχολή και ε, ε, μεταξύ των διαφόρων σχολών στην ίδια χώρα, ώστε είναι δύσκολο να είμαστε σίγουροι πάντα. Και υπάρχει μια δυσπιστία μεταξύ των διαφόρων πανεπιστημίων. Και τα πανεπιστήμια συνέβαλαν για την μικρή επιτυχία του έρασμου, αν και είδα ότι από πέρυσι είχαμε μια σαφή βελτίωση ε, στις ανταλλαγές ε, μέσω του προγράμματος Έρασμος. Πολύ συχνά τα πανεπιστήμια, επειδή δεν έχουν τα διοικητικά μέσα για να συμπληρώσουν τις αιτήσει και τους φακέλους και δεν είναι και καλά ενημερωμένα, πολύ συχνά τα ίδια τα πανεπιστήμια είναι διστακτικά απέναντι στην πρόθεση των φοιτητών τους να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Έρασμος ε, και φοβούνται ότι δεν θα προλάβουν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών τους, οι φοιτητές τους. Ε, αυτό οφείλεται και ε, με τα modules που δίνουν μια ελαστικότητα στην επιλογή και ένα, μια ανοιχτή μεγάλη ελευθερία επιλογή στους ε, φοιτητέ, αλλά θα πρέπει να γίνει καλύτερο συντονισμός ε, και να απαλληλθούν οι διαφορές μεταξύ των χωρών, φυσικά με σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων, αλλά να βρούμε ένα ελάχιστο κοινό παρονομαστή, ένα ελάχιστο κοινό κορμό, ιδιαίτερα στις Χώρε που έχουν πιο επιτακτική νομοθεσία και πιο περιοριστική και που αφήνουν λιγότερη επιλογή στου φοιτητέ. Ε, να γεφυρώσουμε το κενό μεταξύ αυτών των χωρών και των άλλων που είναι πολύ πιο χαλαρέ και αφήνουν μεγαλύτερη ελευθερία επιλογή στου φοιτητέ του. Πάντω, αυτό που είναι κέριο για μα είναι η παράγραφο 6 και ο συνδυασμό με τη διευκόλυνση τη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, γιατί αναφέρεται το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφορών Τακτικών Μονάδων και η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως συγκριτικό εργαλείο. Επίσης, ε, να λάβουμε υπόψη και τις δεξιότητες και όχι μόνο το περιεχόμενο, τις δεξιότητες που προσφέρουν και όχι μόνο το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών. Πολύ φιλόδοξη όλα αυτή η στόχη, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε και ένα εργαλείο για σύγκριση και να ενθαρρύνουμε και τα κράτη-μέλη αλλά και τα πανεπιστήμια να συντάξουν ε, καταλόγους ε, συγκριτικούς, πίνακες σύγκρισης σε ό,τι αφορά την κατανομή των μορίων. Γιατί για συγκρίσιμα μαθήματα μπορούμε να έχουμε 3-4 μόρια στη μια χώρα και 10-12 για το ίδιο μάθημα σε άλλη χώρα ή σε άλλο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι αρνητικό και για τους φοιτητές, αλλά και για την ίδια την ευρωπαϊκή πρόταση και προσέγγιση αυτού του θέματος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για τις προτάσεις. Άλλος κανείς θέλει το λόγο. Δεν ξέρω, ίσως ο κύριος Τάισορ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να υποβάλει κάποια σχόλια τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επιτροπή σα για το ενδιαφέρον που δείχνει. Η εκπαίδευση είναι σημαντικό ζήτημα και δεν μπορούμε να το αφήσουμε στου εκπαιδευτικού. Και χαίρομαι για το ότι η Επιτροπή σα ασχολείται με ναι, αυτό. Οι βουλευτέ θα είδαν βεβαίω πω η Κομισιόν έβγαλε μια ανακοίνωση για τον εξυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και θα είδατε βεβαίω πω συνδέονται οι συστάσει τη ηγήτρια και τη Κομισιόν όσον αφορά τι προτεραιότητε για το μέλλον. Γιατί μαζί με το σημαντικό ρόλο των πανεπιστημίων και λοιπόν ανωτά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σημαντικό είναι να επεκτείνουμε την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, να μειωθεί ο ρυθμός εγκατάλειψης του σχολείου, να προσαρμόσουμε το πώς ε, μπορούμε να εκπληρώσουμε τις ανάγκες των πελατών της ανώτατης εκπαίδευσης με ζητήματα όπως η διάρθρωση που ανέφερε ο κύριος Πρόεδρος. Πρέπει λοιπόν να αυξηθεί η ποιότητα των ε, προγραμμάτων σπουδών και η πτυχή της απασχολησιμότητας και το τι ζητάνε οι εργοδότες ε, από τους ε, πτυχίουχους. Επίσης βεβαίως είναι τα πανεπιστήμια επίσης παιδεία, δημιουργικότητας και έρευνας. Όλα αυτά καλύπτονται στην ανακοίνωση της Κομισιόν. Όσον αφορά την Πολόνια, όπως είπε η ε, Αντιπρόεδρος, πρέπει να γνωρίσουμε πως είχαμε μεγάλη πρόοδο στα 10 χρόνια ύπαρξης ύπαρξη ε, της Μπολόνιας, της διαδικασίας της Τα δύο τρίτα των χωρών ε, που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία έχουν το 90% των προγραμμάτων τους σε αυτή τη διάρθρωση bachelor, master, διδακτορικό και 75% των κύκλων σπουδών χρησιμοποιούν το πρόγραμμα ανταλλαγής διδακτικών μονάδων στις 45 από τις 47 χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία, οπότε πολλά έχουν γίνει δυστυχώς. Και εδώ πέρα έρχομαι σε κάτι που ενδιαφέρει ειδικά την Επιτροπή σας, το 25% των μαθηματών κύκλων σπουδών που ακολουθούν αφορούν τα ρυθμισμένα επαγγέλματα και πάνε υπάγονται άρα στην οδηγία περί επαγγελματικών προσώπων και βεβαίως η Κομισιόν ρώτησε πάρα πολύ εντατικά στη διαβούλευσή τη για τι σχέσει μεταξύ μπολόνια, διαδικασίας Μπολόνιας και επαγγελματικών προσόντων. Είναι δύσκολο να δούμε αυτή τη στιγμή το πώ μπορεί να γίνει αυτό δεδομένη τη άνηση εφαρμογή του ECTS στα κράτη-μέλη. Και πέραν των εκκλήσεων στα κράτη-μέλη και στην Κομισιόν που έχουμε εδώ, θα μπορούσαν να γίνουν και κάποιες εκκλήσεις στα ίδια τα πανεπιστήμια, γιατί αυτά είναι υπεύθυνα για την ύλη και θα γίνουν ακόμη περισσότερο καθώς αυξάνεται η αυτονομία και η ανεξαρτησία τους. Θα υπάρξει επίσης μια έκθεση για την ε, διαδικασία της Μπολόνιας που θα παρουσιαστεί στην διάσκεψη του Βουκουρεστίου τον Απρίλιο του επόμενου έτους και η Κομισιόν συνεισφέρει μέσω του δικτύου Δίκη και ως αποτέλεσμα της εμπλοκής μας ε, η έκθεση αυτή θα είναι πολύ πιο λεπτομερής και άρα ελπίζω να είναι χρήσιμη για το Κοινοβούλιο. Καλώς ορίζουμε λοιπόν τα όσα ακούστηκαν στο σχέδιο αυτό και από τους βουλευτές απόψε και αναμένω την περαιτέρω συνεργασία μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Very much indeed. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για να κλείσει. Μας δώσατε ήδη τις προθεσμίες, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μακλάκεν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για, για τα σχόλιά σας και για τις ιδέες σας και τα σχόλια της Επιτροπής. Πράγματι είναι πολύ δύσκολο με τους περιορισμούς που έχει κανείς να βάλει όλα αυτά μέσα. Προφανώς θα υπάρξει αναφορά στο πρόγραμμα Εράσμους που έχει δώσει τεράστιες εμπειρίες σε τόσους πολλούς φοιτητές και θα υπάρξει μια τροπολογία προς την κατεύθυνση αυτή. Θα ήθελα να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στο ότι μπορεί να συνδέσει την εσωτερική αγορά με την έκθεση αυτή κόμη. Πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε και την κινητικότητα των ερευνητών και πώς να μπορέσουμε να συντονίσουμε τα διάφορα όργανα και να διασφαλίσουμε ένα διάλογο ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στις σχολές, έτσι ώστε να υπάρχουν οι δυνατότητες στους φοιτητές να ταξιδεύουν όχι μόνο για σπουδές αλλά και για μαθητείες. Περιμένω λοιπόν να συνεργαστώ ακόμα περισσότερο με τους ιητές. Ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία είναι 27 Οκτωβρίου και θα ψηφίσουμε στις 22 Νοεμβρίου πράγματι. Να πω επίσης ότι αυτό θα είναι τμήμα των τελευταίων τεσσάρων συνεδριάσεων για φέτος της Επιτροπής. Δεν ξανασυναντιόμαστε μέχρι τις 23 Νοεμβρίου. Κάποιοι από εμά πηγαίνουν στην Τουρκία, στην αποστολή για την Τουρκία, για πολλά ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με την εσωτερική αγορά και την προστασία του καταναλωτή και θα γίνει άλλη μία συνάντηση στις 5 Δεκεμβρίου, η τελευταία. Υπάρχει δυνατότητα συνάντησης και στις 20 Δεκεμβρίου, αλλά θα δούμε αν θα την οργανώσουμε ή όχι. Λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο θέμα. Θα έχουμε μία σύντομη τώρα συνάντηση των εισηγητών. Ευχαριστώ τους, ε, των συντονιστών, συγγνώμη. Έχουμε τώρα να ευχαριστήσω τους, τους εισηγητές και για τις νομοδοτήσεις και για τις εκθέσεις τους. Ευχαριστώ και τους και όλους τις ηγητές. Θα διακόψουμε για λίγα λεπτά έτσι ώστε να μπορέσουν να φύγουν αυτοί που δεν μπορεί να είναι παρόντες στη συνάντηση των συντονιστών και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε.